Good afternoon. Ladies and... Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε όλοι Καλώς ορίσατε σε αυτή τη συνεδρία της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών Προέδρων των Αρμοδίων Επιτροπών. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όσους έρχεστε από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω έναν αριθμό παρατηρητών από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο καθώς και από τα κοινοβούλια του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους εσάς. Επίσης, δεν είναι και κλεισμένο το θηρόν συνεδρίαση και θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα δημοσιογράφων από τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι στις Βρυξέλλες για ορισμένες μέρες. Καλωσορίσατε όλοι εσείς. και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε όλοι τους προσκεκλημένους μας. Καταρχήν, θα ήθελα να καλωσορίσω μεταξύ μας και είναι μεγάλη μας ε, τιμή και ικανοποίηση να καλωσορίσω τον ε, νέο υπατό εκπρόσωπο της ε, Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και την πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπορέλ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. και καθώς ο κύριος ε, Μπορέλ πιέζεται από το χρόνο και θα πρέπει να πετάξει στην Πρατισλάβα αργότερα μέσα στη μέρα, θα ήθελα καταρχήν να δώσω σε αυτόν το λόγο για να παρουσιάσει το σχέδιο δράσης του ως ε, ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος και κατόπιν θα έχουμε χρόνο για τη συζήτηση και θα μου πείτε πότε πρέπει να φύγετε. Έχετε το λόγο κύριε Μπορέλ. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ όλους. plan. Ένα σχέδιο εργασίας είναι κάπως υπερβολή. Αλλά θα μοιραστώ μαζί σας τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εκ νέου εδώ. Είναι πραγματικά η τρίτη μου ημέρα από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως υπαντός εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο. Ε, πήγα στο Παρίσι, στο Κουρτέ Αμβαλίντ, για να ποτίσω φοροτιμή στους Γάλλους ε, στρατιώτες ε, που σκοτώθηκαν στο Σαχέλ στο Μαλί τις προάλλες και μάλιστα παρευρέθηκαν και στη Μαδρίτη στην ανακτήρια συνεδρίαση της διάσκεψης για το κλίμα. Πρόκειται για δύο πολύ συμβολικά γεγονότα στο σημερινό μας κόσμο. Επίσης, συμβολίζουν το έργο που έχουμε να ελοπίσουμε. Σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση του Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήσαμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και την εξωτερική και διεθνή διάσταση αυτής της ε, πολύ σημαντικής πρόκλησης για την Ευρώπη. Κατά την ακρόασή μου εδώ, είπα ότι θα ήθελα να συνεργαστώ σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί είμαι πεπισμένος για το θεμελιώδη ρόλο που θα διαδραματίσετε στο να καταρτήσετε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Όμως, για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να είναι και ενωμένη. Και σήμερα έχουμε πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και δεν μπορούμε να τα αποκρύψουμε όλα αυτά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να οικοδομήσουμε μια κοινή πολιτική υπερβαίνοντας τις δυσκολίες. Θα επικεντρώσω τα εισαγωγικά μου σχόλια σε δύο μέρη. Καταρχήν, τη θέση της Ευρώπη σε ένα πιο ανταγωνιστικό κόσμο και δεύτερον, την ανάγκη και το νόημα αυτής της γεωπολιτικής προσέγγισης. Πρόκειται για μια γεωπολιτική επιτροπή που ανέφερε πολλά και εσύ ήδη η πρόεδρος Φαντερ Λάιεν. Είναι νομίζω σαφές ότι η επιστροφή στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων συμβαίνει ενώ η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική αλεξάρτηση θεωρούσαμε ότι θα τη μειώσει. Όμως αντιθέτως ο στρατιωτικός ανταγωνισμός επανέρχεται πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Και η στρατιωτική μας προσπάθεια θα πρέπει τώρα να αυξήσει και να αυξηθεί, συγγνώμη, και επισωτικά και ποτικά. Και σήμερα είναι μια καλή μέρα να το συζητήσουμε αυτό, καθώς όπως γνωρίζετε σήμερα λαμβάνει χώρα και η συνεδρία του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. και υπάρχουν πολλές διαφωνίες για να το θέσουμε έτσι ή έντονες δηλώσεις για το μέλλον του οργανισμού. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι παρά τον τεράστιο πλούτο και τη δημιουργικότητά μας, η Ευρώπη και μόνο για δημοκρατικούς λόγους θα δει να αποδυναμώνεται η οικονομική της μεγέθυνση τις επόμενες δεκαετίες παγκοσμίω. Επομένως, η ενότητά μας αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωσή μας. Και η άμυνα είναι ένα από τα εργαλεία κλειδιά αυτής της επιβίωσης. Βλέπουμε να επιστρέφουν σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικές πολιτικές. Υπάρχουν ε, διάφορες απειλές ε, που έρχονται από μη κρατικούς φορείς στην περιφέρεια της Ευρώπης ε, και βλέπουμε ε, να, τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ. Οι απειλές ε, προστίθενται. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα σύνολο εργαλείων ευρύτερων, πιο ευέλικτων και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ταχύτατα. Το κλασικό μέσο της διπλωματίας, της soft power όπως αυτό αποκαλούμαστε, εμπόριο, τεχνολογία, επιστήμη γίνεται σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών. Ουσιαστικά τα δύο είδη εξουσίας, soft and hard power, τα δύο είδη ισχύος και δύναμης, αλληλοαναμειγνύονται. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε είναι να αντιδράσουμε συλλογικά στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά θα ε, γίνουμε ουσιαστικά η παιδική χαρά των άλλων. Όλοι εσείς ε, στο έργο σας, στο κοινοβουλευτικό, το βλέπετε αυτό καθημερινά. Οι Ηνωμένε ε, Πολιτείες επιδιώκουν μία μονομερή προσέγγιση προς την Ανατολή περισσότερο, αντιμετωπίζουμε απειλές από την Ανατολή και η Κίνα ε, την ορίζαμε ως οικονομικό εταίρο, αλλά τώρα παρουσιάζεται και ως εχθρός. Ε, υπάρχει Υπάρχουν προκλήσεις που παρουσιάζονται στην Αφρικανική Ήπειρο. Την επόμενη Δευτέρα, στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών, θα ασχοληθούμε με το θέμα της Αφρικής για να προετοιμάσουμε την ε, σύνοδο κορφής με τις χώρες της Αφρικής και η πρόεδρος η Ουρσουλα von der θα επισκεφθεί σύντομα την Αφρική. Η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, οι βρεδικές απειλές, ε, εκστρατείες παραπληροφόρησης, όλες αυτές οι νέες απειλές δεν είναι τα είδη των απειλών που προσπαθούσαμε να απαντήσουμε εφαρμόζοντας το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ παραμένει το βασικό μέσο εδαφικής άμυνας για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και νέες απειλές που χρήζουν συγκεκριμένης απάντησης. Και αυτή η συγκεκριμένη απάντηση θα πρέπει να ενεργοποιήσει τις ενεργές μας. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πριν να γίνουν οξία. Χρειαζόμαστε μια ε, στρατηγική νοοτροπία προκειμένου να συμφωνούμε περισσότερο. Και σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούμε στο να δρούμε ταχύτερα όταν πρέπει. Και τέλος, καθώς απευθύνομαι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο προπολογισμό για την εξωτερική δράση που να μας δίνει τα μέσα να προωθήσουμε την παγκόσμια παρουσία μας και να απαντήσουμε ταχύτατα σε καταστάσεις κρίσης. Η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ε, είπε σήμερα στο Παρίσι ότι αναμένει 30% αύξηση στη χρηματοδότηση για τις εξωτερικές πολιτικές. Και είμαι σίγουρη ότι εσείς θα την υποστηρίξετε ακόμη και αν ένα 30% μάλλον ε, θεωρείται υπερβολικό, δηλαδή όχι υπερβολικό, εντάξει είναι δύσκολο να το πετύχουμε εννοώ. Δεύτερον, η ανάγκη για μια γεωπολιτική προσέγγιση και τι σημαίνει αυτό. Όλοι επαναλαμβάνουν την πρόταση της κυρίας Φοντερ Λάιεν, ότι πρόκειται για μια γεωπολιτική επιτροπή. Επίσης, ακούσαμε την έκκληση του Πρόεδρου Μακρόν ε, στην συνέντευξή του, ε, στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με τον Πρόεδρο ε, Τραμπ. Τα σχόλιά του για το ΝΑΤΟ προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή και πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. Η συνάντηση των αρχηγών κρατών στο Λονδίνο μόλις έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, αν και είναι σαφές ότι σημαντικά θέματα μεταξύ των συμμάχων πρέπει να συστηθούν περαιτέρω. Νομίζω ότι πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Ειλικρινά, πρέπει να γίνει συζήτηση μεταξύ μας. Το ΝΑΤΟ έχει σημαντικά από όλα μάλλον τα σημαντικά πολιτικά project έχει υποστεί και κάποιες κρίσεις κατά τη διάρκεια τη ύπαρξή του. Αυτή δεν είναι η πρώτη και έχει καταφέρει να τις ξεπεράσει επιτυχώς. Κατά την ε, δική μας εμπειρία, στην πραγματικότητα, οι κρίσεις ε, συχνά οδηγούν σε ενδυνάμωση. Και η σημερινή κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προχωρεί στη δική της ε, ανάπτυξη ως ένας διεθνής πρωταγωνιστής ασφάλειας και να αρχίζει να σκέφτεται στρατηγικά τον εαυτό της ως γεωπολιτική δύναμη. Διαφορετικά το μέλλον μας θα αποφασίζεται από άλλους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να αντιμετωπίζουμε σοβαρά το θέμα της οικοδόμησης ολοκληρωμένης ε, εξωτερικής ε, πολιτικής. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνοχής ε, των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Είναι μεγάλη πρόκληση. Καταλαβαίνετε να διασφαλίσω τη συνοχή των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει το έργο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Κομισιόν των Κρατών Μελών να το ευθυγραμμίσουμε με ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Και επαναλαμβάνω, ζούμε σε ένα γεωπολιτικό κόσμο, είμαστε, έχουμε μεγάλους παίκτες, τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, αλλά και την Τουρκία μεταξύ άλλων. Όλοι αυτοί δρούν με γεωπολιτικό τρόπο. Τα ανοιχτά θέματα θα μας οδηγήσουν στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη της ισχύω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα είπαν ότι δεν υποστηρίζουν το φόρο για τους μεγάλους γίγαντες της ψηφιακής οικονομίας και απειλούν με αντίμετρα κατά των χωρών που θεθετήσουν αυτά τα μέτρα. Λιβύη. Η Λιβύη είναι ένα καλό παράδειγμα. Θέλουμε να συζητήσουμε για τη Λιβύη. Είναι ακριβώς απέναντί μας στη Μεσόγειο. Η αστάθεια στη Λιβύη απειλεί άμεσα τη δική μας ασφάλεια και θέτει προκλήσεις απέναντι στις αξίε μα ε, σε σχέση με το μεταναστευτικό και του ετούντε άσυλο. Είναι άμεσος γειτονά μα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετική θέση και να συνεργαστεί με περιφερειακούς παίκτες και την υποστήριξη του ΟΗΕ για να βρεθεί μια πολιτική λύση για αυτή την αποτυχημένη χώρα. Αυτό το λέμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει συμβεί η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται και έχει πολλές αλλαγές και παρεμβαίνουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις διμερείς δράσεις γιατί πυροδοτούν περαιτέρω τη σύραξη στη Λιβύη και αυξάνουν την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόσπατη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης σε σχέση με τα ύδατα στη Μεσόγειο και ακόμη δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, αλλά έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες στην Ελλάδα και μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας πριν πετάξει στο Λονδίνο. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα. Εμείς είμαστε μεγάλη διπλωματική δύναμη. Είμαστε και οικονομική υπερδύναμη. Η εμπορική μας πολιτική είναι επιτυχής παρά την κριτική εμείς ε, έχουμε οικοδομήσει και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα δίκτυο εμπορικών συμφωνιών και θα θέλουμε να έχουμε την προϋπόθεση να είναι βιώσιμο ως προς την ανάπτυξη. Στις διαπραγματεύσεις μας θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, όλο και περισσότερο. Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ε, ιδίως με την ΠΕΣΚΟ και το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Τεμείο που θα πρέπει να συζητήσετε υπό τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, θα προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ ε, είμαι πρόεδρος του κλάστερ για τις εξωτερικές σχέσεις. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τους κανόνες της διαδικασίας στο σώμα, δηλαδή για το πώς θα εργαστούμε και έχω την ευθύνη κάθε εβδομάδα να παρουσιάζω την κατάσταση των διεθνών προβλημάτων ε, και να προεδρεύω μιας ε, ομάδας επιτρόπων που σχετίζονται πιο άμεσα με τις εξωτερικές πολιτικές. Αν και η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση δεν είναι μεταξύ αυτών και είναι μέρος των πιο σημαντικών διεθνών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να δώσουμε ένα πρώτο παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ας μιλήσουμε για το ποιο θέτει τους κανόνες. Αυτός που θέτει τους κανόνες ε, θα εξουσιάσει και τον κόσμο. Είμαστε σε ένα ιδεολογικό πόλεμο. σχετικά με τους κανόνες και με την ιστορία που θα φυγηθούμε στους πολίτες. Και τι θα σημαίνει αυτό για το πώς κατανοούμε τον κόσμο. Δείτε το σχάρι τι σημαίνει με τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Είναι το αίμα της νέας οικονομίας τα δεδομένα. Σύμφωνα με κάποιον η συνολική αξία των δεδομένων μάλλον της οικονομίας ε, που κινείται από τα δεδομένα είναι μεγαλύτερη από την αξία του παγκόσμιου εμπορίου σε πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν οι κανόνες για τα δεδομένα έχουν τόση σημασία όσο οι κανόνες στον τομέα της ενέργειας. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, οι κανόνες υπονοούν ότι τα δεδομένα ανήκουν στις εταιρείες του τεχνολογικού τομέα ή στις τεχνολογικές πλατφόρμες. Στην Κίνα τα δεδομένα ανήκουν στο κράτος. Στην Ευρώπη τα δεδομένα ανήκουν στα άτομα. Ποιο μοντέλο θα κερδίσει τελικά, οι εταιρείε, το κράτος ή τα άτομα, δηλαδή η κοινωνία. Εμείς στην Ευρώπη δικαίως είμαστε περήφανοι για το μοντέλο μας σχετικά με την οργάνωση των κοινωνιών και των οικονομιών μας. Δεν θέλω να θριαμβολογώ αλλά έχουμε ένα αληθινό μείγμα οικονομίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τη δεκαετία του 90 πιστεύαμε ότι θα είχαμε παγκόσμια πρόκληση σύγκλησης γύρω από τις έννοιες αυτές. Αλλά δεν συνέβη, το ξέρουμε τώρα. Αντιθέτως, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών συστημάτων η Κίνα είναι συστημικός ε, αντίπαλος ε, και αν το πούμε αυτό τι εννοούμε. Τι σημαίνει ο όρος σύστημα συστημικός αντίπαλος. Σημαίνει ότι υπάρχει αντιπαλότητα σε σχέση με τα συστήματα και δεν είναι προφανές ότι μια ομάδα χωρών που σήμερα αποτελεί κάτω από το 90% του παγκοσμίου πληθυσμού θα υπερισχύσει εκτός και επανέρχομαι στην αρχή της παρέμβασής μου εκτός και αν δράσουμε όλοι μαζί. Ε, εμείς γιορτάσαμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ήμουν στο Βερολίνο και πολλοί πίστευαν ε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ε, στο σύστημα της ελεύθερης δημοκρατίας, στην οικονομία της αγοράς. Αυτό είναι το τέλος της ιστορίας, κάποιοι έλεγαν. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει. Το σοβιετικό σύστημα δεν ήταν καλύτερη εναλλακτική για την ευμερία των λαών, όπως πολλοί εξημών γνωρίζετε πολύ καλά. Στην Κίνα όμως, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια, υλοποιώντα μία από τις πιο θεαματικές μεταμορφώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, η Αφρική θα έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους παραπάνω. Χθε ήμουν με τον Τζέφρι Σάντς και μιλούσαμε για τη δημογραφική έκρηξη της Αφρικής και πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε, τα αριθμητικά στοιχεία που έρχονται, χωρίς κανείς να μπορεί να τα διαχειριστεί. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε την Αφρική μόνο μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονό ότι η δημογραφική ανισορροπία και οι ανισότητες του πλούτου μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου θα αυξηθούν ιδιαίτερα. Μόνο αν δράσουμε από κοινού μπορούμε να αποτελέσουμε εταίρο της Αφρικής και μόνο αν δράσουμε από κοινού μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση με την Κίνα προσέγγιση μας θα βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως δεν είναι σαφές ότι οι εταίροι μας θα έχουν τον ίδιο στόχο. Επομένως θα πρέπει να επιμείνουμε στο τι σημαίνει αυτή η ε, νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Green New Deal που συζητήθηκε χθε στην Κομισιόν και στη Μαδρίτη στη διάσκεψη για το κλίμα. Συνολικά, η φύση της ε, εξωτερικής πολιτικής αλλάζει. Η εξωτερική πολιτική δεν ε, ήταν ε, ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η εξωτερική πολιτική δεν αφορά μόνο τη διπλωματία, καλύπτει κάθε πτυχή της βιομηχανικής, τεχνολογικής, γεωπολιτικής επανάστασης που πλησιάζει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε μεγάλο επίπεδο, σε συνολικό επίπεδο, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Να πω και κάτι για κάποιες γεωγραφικές προσεγγίσεις. Καταρχήν, Δυτικά Βαλκάνια. Ήδη και αυτά ήταν στις ειδήσει και υπήρξε μεγάλη απογοήτευση στα Βαλκάνια σχετικά με την ε, μη δυνατότητα την άρνηση τη συνέχιση της διαδικασία της διεύρυνση. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων. Όπω είπα στην ακρόασή μου, θα ήθελα να μεταβώ σύντομα στο Κωσυφοπαίδιο και στη Σερβία, όπου στο Κωσυφοπαίδιο δεν υπάρχει ακόμα κυβέρνηση και δεν είναι χρήσιμο να μεταβώ πριν ε, να αναλάβει καινούργια κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν δεν ε, μπορώ να υλοποιήσω την υποσχέση που έδωσα την πρώτη μου επίσκεψη θα είναι στο Κωσυφοπέδιο, θα πάω στην Πρετισλάβα που είναι εκεί κοντά, γιατί σήμερα φιλοξενεί τις συνεδρίες του ΑΣΕ και θα συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας αλλά και όλων των άλλων χωρών της Ανατολής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία καθώς και τη Γεωργία και την ε, Δημοκρατία της Μολδαβίας. Όπως είπα, θα πρέπει να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο στο να βοηθήσουμε να ξαναοικοδομηθεί το κράτος της Λιβύης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους. Θα πρέπει να έχουμε μια συντολική προσέγγιση στις πολλαπλές σειράξεις στον κόλπο. Την επόμενη εβδομάδα θα προεδρεύσουμε την συνεδρίαση για την πυρηνική συμφωνία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει εντελώς ακυρωθεί και σε αυτό το πνεύμα θα συναντήσουμε, θα συνεδριάσουμε μάλιστα στη Μεκτή Επιτροπή αύριο και την Παρασκευή. Και τέλος, δύο λόγια για το Σαχέλ. Απλώς για να ποτίσω φοροτιμή στους Γάλλους στρατιώτες που σκοτώθηκαν εκεί. Εκεί η τάση παραμένει αρνητική. Ήμουν στο Παρίσι για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στη Γαλλία για τις απώλειες του στρατού και θέλω να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε συλλογικές προσπάθειες να αναλαμβάνουμε στο Σαχέλ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιες λίγες ευρωπαϊκές χώρες να φέρουν το άχθος ή να διασφαλίζουν την ασφάλεια αυτού σε αυτό το μεγάλο μέρος της Αφρικής, ενώ αυξάνεται η δημογραφική βόμβα και ενώ τα κράτη δεν μπορούν να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δεσμευόμαστε ε, και να συμμετέχουμε στο τι συμβαίνει σε αυτό το τμήμα του κόσμου, γιατί πολλές από τις απειλές εποάζονται εκεί. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Περιμένω να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων για αυτά και άλλα ζητήματα. Σήμερα δημοσιεύσαμε και μια ανακοίνωση, ίσως την πρώτη, ένα ανακοινωθέν τύπου, την πρώτη της αιτίας μου και αναφερόμαστε στη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που ανησυχεί πάρα πολύ την Ελλάδα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία στη συνάντηση στην Πρατισλάβα απόψε και αύριο. Είμαι στη διάθεσή σας για να έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Γιατί πιστεύω πρέπει τα πράγματα να τα λέμε ξεκάθαρα μεταξύ μας. Υπάρχουν πολλές διαφορές, πολλές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ο μόνος τρόπος να τις ξεπεράσουμε είναι αν τις εξηγήσουμε για να καταλάβουμε τους λόγους που έχει η κάθε χώρα απέναντι σε συγκεκριμένα προβλήματα. Και ξέρω ότι αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις βασίζονται στην ε, ιστορία μας, που είναι βαθιά ε, ριζωμένη. Έχει βαθιές ρίζες ε, σε αιώνες πίσω. Αλλά αν θέλουμε να σφυρατήσουμε ένα κοινό μέλλον, θα πρέπει να υπερβούμε αυτές τις διαφορές και να οικοδομήσουμε μια κοινή ιστορία για την επιβίωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε, Λέω ο Πρόεδρος τον Αντιπρόεδρο και είπα το εκπρόσωπο Μπορέλ, συνάδελφοι, τα πράγματα έχουν ως εξή. Έχει 50 λεπτά στη διάθεσή του ο κ. Μπορέλ. Έχω πολλά αιτήματα από ομιλητές και πρέπει να σεβαστώ γεωγραφική κατανομή, πολιτικές ομάδες, ισότητα φύλων και άλλα πολλά. Mission impossible είναι, λέει ο πρόεδρος. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσω το λόγο στους φιλοξενουμένους μα από τα κράτη-μέλη και σίγουρα σε κάποια μέλη. Κύριε Μπορέλ, σταματήστε μας αν νομίζετε ότι έχετε σωρεύσει αρκετές ερωτήσεις. Ωραία, θα ακούσουμε κάποιες μαζί και επομένως εσείς έχετε την ευθύνη, οπότε θα μας σταματήσετε να μην ακούσετε άλλες ερωτήσεις. Πρώτος ομιλητής, λοιπόν, Έχουν διανεμηθεί και κάρτες ε, στους φιλοξενούμενους. Και σας παρακαλώ ένα λεπτό, ενάμιση, έχω και το σφυράκι μου εδώ. Λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κόβαξ από την Κροατία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μπορώ να παραμείνω άνδρας παρά τα της ισότητας των φίλων και να μην αλλάξω το φίλο μου. Δηλαδή, χαίρομαι, λέει ο μιλητής. Ε, χαιρετώ θερμός τον αντιπρόεδρο και είπα το εκπρόσωπο. Άκουσα προσεκτικά την εισήγησή του και συμφωνώ με τον κύριο Μπορέλ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικονομική και πολιτική δύναμη και θα πρέπει, μάλλον οικονομική δύναμη και πρέπει να γίνουμε και πολιτική δύναμη και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διαδραματίσουμε ένα ρόλο διεθνώς. Πρέπει δηλαδή να δείξουμε στον κόσμο και στον εαυτόν μας ότι εμείς φροντίζουμε τα θέματα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και με την υποστήριξή σας του χρόνου ελπίζω να έχουμε μια απόφαση για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόβατς. Για το ΕΛΚ, η κυρία Σόφκο. Εδώ είμαι, κύριε Μπορέλ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά για χάρη των συναδέλφων. Όπως είπε και ο συνάδελφος από, την, από το Κοινοβούλιο μας, ε, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή που μας ενδιαφέρει πολύ. Είχαμε τη στρατηγική, είχαμε τα θέματα ασφάλειας και σταθερότητας θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνετε μια επίσκεψη ώστε να διαβάσετε και ένα συμβολικό μήνυμα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας για εσάς γιατί είναι ένας κοινό παρανομαστής επί του οποίου μπορούμε να οικοδομήσουμε την κοινή μας εξωτερική πολιτική στο μέλλον. Και η ασφάλεια είναι σημαντικό διακύβευμα, μια και είμαστε όμοιροι πλέον της Τουρκίας ε, για τους εκατομμύρια πρόσφυγες ε, που μπορεί να εξαπολύσει αν δεν φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Και το αίτημά μου θα ήταν να παρακολουθήσετε την σύσταση, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τις χώρες αυτές και να το θεωρήσετε προσωπική σας αποστολή ότι η ειρήνη και η ασφάλεια θα είναι ύψης της προτεραιότητας τα νότια-ανατολικά σύνορα και στην νοτιοανατολική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε το ρόλο που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουτιέρες από την Ισπανία, από, την, ε, από το Κοινοβούλιο, το Ισπανικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ισπανικά αν μου επιτρέπετε. Χαιρετίζω και εγώ τον κύριο Μπορέλ. Εμείς είμαστε υπερήφανοι Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Είμασταν στο 25, σήμερα είμαστε στο 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είμασταν στο 25, σύντομα θα είμαστε στο 16% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να λάβουμε αποφάσεις ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί με διάφορες χώρες στον κόσμο. Πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό υπάρχει θεσμική πολιτική κρίση στην Νότιο Αμερική, τι ρόλο πρέπει να δεματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί και η Ισπανία ειδικά ως άμεση γέφυρα με την Νότιο Αμερική. Επίσης η μεταναστευτική πολιτική και οι μεγάλες συμφωνίες. Έχουμε συμφωνίες ποσοστώσεων. Ποια είναι η ισορροπία θεωρείτε εσείς ως υπεύθυνο της πολιτικής της ασφαλείας ε, των ελέγχων των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής. Στο Σαχέλ ιδιαίτερα ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που έχουμε θέσει τον εαυτό μας εκεί, ιδιαίτερα για την μεταναστευτική πολιτική. Συγχαρητήρια και πάλι ο πλευρά μου ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέω ο Πρόεδρος. SND, ο κύριος Πίτσουλα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Μπορέλ, πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θερμά συγχαρητήρια και πολύ καλή επιτυχία για όλες τις ε, προσπάθειές σας ως Αντιπροέδρος και είπατε ως εκπρόσωπος. Στη δήλωση προθέσεών σας είπατε ρεαλισμός και ενότητα ως κατευθυντήριες αξίες ε, για να καθοδηγήσουμε την ε, πολιτική ασφαλείας και την εξωτερική πολιτική που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να δρούμε ως ευφυής δύναμη συντονισμένα μεταξύ των θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Αυτό βέβαια θα ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή ως προς το πώς λειτουργούμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ ε, η εγγύηση ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ για την ασφαλειά μας, αλλά πολύ σημαντικά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει την ε, δυσαρέσκειά τους και τη διαφωνία τους για το μέλλον του ΝΑΤΟ. οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται να υποχωρούν από το σύστημα της πολυμερίας και η ερώτησή μου είναι ως ύπατος εκπρόσωπος εσείς πώς θεωρείτε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί ένας απεικοδομητικός διάλογος με τα κράτη-μέλη ώστε να έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες δυναμικό ασφαλείας, ετοιμότητας και προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Νίνο. Άλλη μία θέλουμε να ακούσουμε. Ωραία από η κυρία Γκρεγκότσιτς από τη Σλοβενία παρακαλώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη Σλοβενία συμμεριζόμαστε το όραμα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας υπεύθυνο ε, παγκόσμιος παίκτη δύναμη και μπορούμε να έχουμε περισσότερη επιρροή με συντονισμένες δράσεις στο παγκόσμιο σκηνικό δεδομένων των ταχύτατων αλλαγών που διενεργούνται βλέπουμε ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ισχυρός ε, συνεργάτης ε, του παγκόσμιου συστήματος πολυμερίας και, για, και στη συνεργασία σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά υβριδικές απειλές. Οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών της Στι σχέσεις του με τρίτε χώρε πρέπει να, είναι, να έχουν μια ομοιογένεια, να, ε, να είναι συντονισμένε και να είναι προδραστικέ. Θα πρέπει να εστιαζόμαστε στην ειρήνη, την ασφάλεια, το κράτο δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Εμεί στη Σλοβενία οπωσδήποτε θα, είμαστε, θα εξεκολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ασφάλεια, ειρήνη και πολιτική σταθερότητα στην γειτονιά μα, με ιδιαίτερη εστίαση βεβαίως στα Δυτικά Βαλκάνια η ιστορία μας διδάσκει ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή με πολλά ακόμα άλλη τα προβλήματα. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή προοπτική είναι λίγο πολύ η πρόθεση και το όνειρο όλων των χωρών της περιοχής αυτής. Πρέπει και εμείς να είμαστε αξιόπαστοι, πιστεύω. Ευχαριστώ κύριο Μπορέλ για να απαντήσει στον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από τα ερωτήματα αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω ακράδαντα πως δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρέπει να παραμείνει στην προτεραιότητα. Το θέμα της διεύρυνσης ήγηρε πρόσφατα κάποια ερωτήματα, το λιγότερο που μπορώ να, που μπορώ να πω. Όμως, μακροπρόθεσμα ή μέσο πρόθεσμα, νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να προετοιμάσουμε τη διάσκεψη κορυφής του Μαΐου του 2020 για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επικροτικής Προεδρίας στο Ζάγκρεπ. Αυτή θα είναι μια καμπή, μια κρίσιμη χρονική στιγμή και τότε θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Στο μεταξύ, νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί η όθηση ε, που έχουμε και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα κρατη ώστε να γίνει αντιληπτό πώς δεν μπορούμε να κλείσουμε ή να ακυρώσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των εν λόγω χωρών. Δεν καταφέραμε να αποτύχουμε τον πόλεμο της Ιουκοσλαβίας. που είχε σχεδόν 150.000 θύματα. Αυτό ήταν μια μεγάλη τραγωδία και κληροδότησε διχασμούς, φτώχεια, εθνοτικούς και εθνικιστικούς αγώνες. Η Ευρώπη είναι η μόνη η οποία μπορεί να προσφέρει λύση σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι στο Συμβούλιο αυτό το ζήτημα θα πρέπει και πάλι να συζητηθεί μέχρι τη συνεδρίαση του Ζάγκρεπα που δικής μου πλευράς μπορώ να σας διαβεβαιώσω την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς αυτό και νομίζω ότι απαντώ με αυτά τουλάχιστον δύο-τρία από τα ερωτήματα. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε το ΝΑΤΟ. Τι γίνεται σήμερα με το ΝΑΤΟ. πώς να το πω, έχουμε τρία-τέσσερα προβλήματα σε διαφορά το ΝΑΤΟ και τη σχέση με ταξί Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Πρώτον, η αντίληψη που υπάρχει πως ε, την είπα την τις είπατε σε ενδιαφέρουν περισσότερο οι ασιατικές χώρες και όχι η Ευρώπη. Αυτό είναι μια αντίληψη της πραγματικότητας, δεν είναι η πραγματικότητα ότι υπάρχει αυτό το σύνορο που είναι ειρηνικό ε, και ότι δεν είναι ε, η Ευρώπη σημαντική για τη ΣΥΠΑ, αλλά η Ασία είναι πολύ σημαντικότερη. Δεύτερο, ε, κάποια συνέπεια, αν θέλετε, στη στάση της Αμερικής απέναντι στη Συρία και τη Λιβύη. Και το έχουμε επικρίνει το θέμα αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε τη στάση αυτή. Τρίτον, το ότι οι ε, δρούν και κινούνται με βάση τα οικονομικά του συμφέροντα. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία οριοθετούν ε, και την ε, θέση της Ευρώπης ότι αφορά το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως, το είπα και στην ακρόασή μου και συνεχίζω να το λέω και να το υποστηρίζω, είναι το βασικό αμυντικό πλαίσιο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τον ΝΑΤΟ ξεπερνώντας τις δυσκολίες αυτές ε, και τις διαφορές αυτές. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναπτυχθούν συμπληρωματικές δυνατότητες από εμάς τους Ευρωπαίους για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα άμεσα προβλήματα. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Όταν φύγουν οι Βρετανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν, εφόσον δηλαδή αποχωρήσουν το 80% των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα ε, προσφέρεται από μη ευρωπαϊκές χώρες. Το 20% μόνο δηλαδή θα χρηματοδοτούμε εμείς των, των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Είμαστε δηλαδή ένα κομμάτι, όχι όμως το σημαντικότερο. Και έχουμε προβλήματα στην άμεση γειτονία που δεν μπορούμε να επιλύσουμε επικαλούμε το άρθρο 5. Και αυτή η αντίληψη για τη ΣΥΠΑ ότι έχει στρέψει ο ενδιαφέρον προ την Ασία, έλλειψη συνέπειε ό,τι αφορά τη Συρία και τον κόλπο επίσης και η πολιτική που ε, βασίζεται στα εθνικά οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτά όλα, όπως είπα, επηρεάζουν ε, την άποψή μας για ε, τη συμμαχία και το ρόλο της. Και προσθέτω τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της Τουρκίας, αν δείτε τις δράσεις της στη Συρία και νομίζω ότι είναι κατανοητές οι ανησυχίες μας. Αλλά μην πιστεύετε ότι αυτή είναι η πρώτη κρίση στο ΝΑΤΟ. Κατά το παρελθόν ήταν πολλές αποκλίνουσες από, 50, από το 56, από την επιχείρηση του Σουέζ, από τους Γάλλους και τους Βρετανούς. Ε, το Κιπούρ, τη Λιβύη το 86, το Ιράκ το 2003 και τη Συρία. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε αυτά τα οποία μας ενώνουν ότι για την Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους το ΝΑΤΟ είναι το βασικό πλαίσιο της συλλογικής μας άμυνας. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. Ακούστε, δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα θα λυθεί με συνοριακού ελέγχου και μόνο. Φυσικά και πρέπει να ανασφαλεί τα σύνορα. Αν ένα κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ε, τα σύνορά του, δεν είναι πλέον κράτος. Άρα ο έλεγχος των σύνορων είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, είναι απαραίτητο αν θέλουμε να νιώθουν ασφαλείς οι πολίτες μας και να είναι ασφαλείς οι πολίτες μας, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Δεν θα ανακόψουμε το μεταναστευτικό ρεύμα αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή του, εκεί που ε, δημιουργείται, όχι εκεί που εκδηλώνεται και γι' αυτό απαιτούνται συμφωνίες εταιρική σχέσης για την ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών. Απαιτούνται συμφωνίες προκειμένου να μπορούν να γυρίσουν πίσω οι παράτυποι μετανάστες να επιστραφούν ταυτόχρονα, να παρασχεθεί άσυλο στους ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται. Η μεταναστευτική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή την Παρασκευή δύο συνάδελφοί μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταβούν στην Άγκυρα για να συζητήσουν με τις τουρκικές αρχές τι θα γίνει με τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στι ελληνικέ ακτές. Δεν είναι πλέον Σύριοι ε, που φεύγουν από τον πόλεμο, αλλά άνθρωποι που έρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, που μπορεί ίσως να προτρέχουν ε, των συνεπειών μια συμφωνία ε, ειρηνευτική με τους Ταλιμπάν. Και το τελευταίο που θα σχολιάσω είναι το ερώτημα για τη Λατινική Αμερική. Και αν μου επιτρέψετε, θα απαντήσω για τη Λατινική Αμερική στα Ισπανικά. Δεν θα ήταν ε, και τόσο δόκιμο να μιλάω στα γαλλικά ή στα αγγλικά για τη Λατινική Αμερική. Ιδίω εφόσον απευθύνομαι και σε Ισπανό συνάδελφο. Αλλά από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, η Λατινική Αμερική πραγματικά πλέον ε, βρίσκεται σε πολύ πιο θερμή κατάσταση. Ε, ήταν το πρόβλημα τότε η Βενεζουέλα και η Κούβα όταν ήρθαν τελευταία φορά. Τώρα έχουμε πάει στη Χιλή, στο Μεξικό. Ε, η μία χώρα μετά την άλλη δηλαδή φλέγεται αν μπορώ να το πω έτσι. Ε, πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική ανατάραχη επικράτη σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και αυτό δεν είναι συνέπεια μόνο των ογκούμενων ανισοτήτων του γεγονότος ότι η δημοκρατία δεν μπόρεσε να αποφύγει τις ανισότητες αυτές ε, στη δεκαετία ε, πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αντιδραστική μάζα και με, το πιο, με μια σπίθα προκαλείται φωτιά. Και έχουμε πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα, πολιτικές αντιπαραθέσεις ε. Τα λέω ε, και δεν τα λέω γιατί είμαι Ισπανός, ε, αλλά γιατί η Ευρώπη πραγματικά πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη προσοχή ε, στη Λατινική Αμερική. Γιατί μέχρι τώρα φαινόταν ότι το μόνο πρόβλημα που, ήταν, που υπήρχε ήταν η Κούβα. Δεν είναι όμως ουσιαστικά το σημαντικότερο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τη Βολιβία, τον Ισημερινό, τη Βενεζουέλα, τη Χιλή και την Κολομβία ο στρατός ξανακατεβαίνει στους δρόμους. Είναι φρικτές οι εικόνες, συνολικά στη Λατινική Αμερική. Ε, έχουμε θανάτους από πυρά, από σφαίρες. Αυτό δεν μπορεί να αφήσει αδρανή και αδιάφορη την Ευρώπη. Νομίζω κάλυψα τις ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο κάποια λεπτά παραπάνω, αγαπητέ Πρόεδρε. Ναι, δεύτερος γύρος, κύριε Μπορέλ, αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε, ωραία. Λοιπόν, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Φων Κραμών. Ευχαριστώ πολύ. Καθώς ήδη αναφέρατε το θέμα του κοσυφοπεδίου, και μπορεί η μεταβασή σας να ελοπιθεί μόνο αφού έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα αναφερθώ σε άλλα δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, αν δούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, θα έχουμε και συνάντηση την επόμενη Δευτέρα ε, και δεν είμαστε μέρος αυτού του φορμά, αλλά ε, θέλουμε να έχουμε, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μια στρατηγική απεύθυνση στην Ουκρανία. Ποια είναι η πρότασή σας για τους Ουκρανούς, για τους Ρώσους, αλλά και για τους Γάλλους και για τους Γερμανούς. Ε, ποια θα μπορούσε να είναι η καταληκτική βιώσιμη λύση. Και δεύτερη ερώτηση. Η ρωσική επιρροή όχι μόνο σε μια γειτονική χώρα, αλλά και στα δικά μας κρατη και επίσης και στη δική σας ε, περιοχή, στην Καταλωνία, ε, στην Ιταλία, στο Brexit, έχουν ανακατευτεί οι Ρώσοι. Ποια είναι τα μηνύματα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να αντιδράσει απέναντι στη ρωσική επιρροή. Ευχαριστώ. Από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο κύριος Λογκλέ από τη Γαλλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πατέ, εκπρόσωπα, ενώ 13 ε, Γάλλοι στρατιώτες από την επιχείρηση Μπαρκάν ε, δολοφονήθηκαν στο Μαλί την περασμένη εβδομάδα. Να υπογραμμίσω ότι η ασφάλεια ολόκληρης ε, της Ευρώπης είναι αντικείμενο υπεράσπισης από τη Γαλλία και η παρουσία σας τη Δευτέρα εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Η ασφαλειά μας είναι ένα κοινό αγαθό, η σταθερότητα του Σαχέλ αφορά και τη σταθερότητα του Μαγκρέβ και της ε, νότιας όχθης της Μεσογείου. Είναι στρατηγική προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, τόπου, η Γαλλία δεν δρά της και έχουμε την υποστήριξη της ε, αποστολής UTM Μαλή και πολλών κρατών μελών ε, είτε από μόνα τους είτε εντό τη μηνουσμά του ΟΗΕ. Φυσικά θα πρέπει όμως να πάμε και πιο μακριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέγιστο ρόλο να παίξει στο πλαίσιο της ε, παγκόσμιας προσέγγισης ε, που δίνει και μεγάλη προστιθέμενη αξία και η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγική για τη διακυβέρνηση, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Ποιο ρόλο θέλει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να προωθήσει τον πολιτικό διάλογο στις χώρες του Σαχέλ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία τελική ερώτηση. Ισπανός συνάδελφος. Και είμαι τόσο ανοιχτό προς Ισπανίδα συνάδελφος, η κυρία Βιγιαλουέβα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Μπορέλ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και καλή τύχη στην, στα νέα σας καθήκοντα. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Καταρχήν, αν θα μπορούσατε να μας πείτε τι σημαίνει η ανεξαρτησία και η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Επιτροπή μας ε, έχουμε πάρα πολλά έγγραφα της κυρίας Μογκερίνη που μιλούσε για τα θέματα αυτά και για την αναγκαιότητα του πολυμερισμού και πώς σκέφτεστε να τελειοποιήσετε με δικές μας δράσεις, με ευέλικτες συμμαχίες, με το διάλογο που χρειάζεται με τη Ρωσία και την Κίνα, με την πρόθεση της ειρήνης και εφαρμόζοντα την κοινή θέση για την πώληση των όπλων, ε, περβαίνοντας ε, την σημερινή φάση εξάρτησης από τον ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, Εκτιμάμε το σχόλιο που κάνατε σε σχέση με την Ελληνική Αμερική και συμφωνούμε. Είναι σημαντικό να μην κοιτάει από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διακυβεύεται η δημοκρατία στην Ήπειρο με πραξικοπήματα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδικάσει αυτά τα πραξικοπήματα, να προωθήσει τη διαμεσολάβηση, να αποφύγει την αυτοδιακηρύξει και να αποφύγουμε την καταστολή των διαδηλώσεων στη Λατινική Αμερική. Εσεί για οικονομικέ ε, δράσει που να βασίζονται στην ανάπτυξη. Εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βασίζονται και σε βασισμό των εργατικών δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και τη αμοιβαία ανάπτυξη και φυσικά να θέσουμε τέλο στου φορολογικού παραδείσου. Και τέλο για την σχέση σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε και στην ακρόασή σας και σήμερα εδώ. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό στο Κοινοβούλιο να υποστηρίζετε το Ευρωπαϊκό Όργανο που έχει το μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα προκειμένου να υπάρξει μια πολύ σημαντική πολιτική και θέλουμε να ακούσουμε τις δεσμεύσεις σας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πολλές απόψεις μαζί σας. Ευχαριστώ. Gracias, señor. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπορέλ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γαλλικά την ερώτηση <clears throat> για το Σαχέλ. Ε, είναι προφανές ότι δεν, είναι αρκετά αυτά που κάνουμε. Βλέποντας το εύρος της περιοχής με πέντε χώρες, ότι τα σύνορα δεν είναι παρά νοητές γραμμές στο χάρτη που δεν υφίστανται στην πραγματικότητα στο έδαφος, βλέποντας την προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη ότι δεν βελτιώνται τα πράγματα. Στο Μαλή ο πρόεδρος, παλαιός φίλος, είχαμε συζητήσει και χθε μαζί του και με τον πρόεδρο του Μπουρκίνα Φάσο, εμείς με τα δικά μας μόνον μέσα δεν μπορούμε να καλύψουμε την επικράτεια, το έδαφος. Γιατί στο Σαχέλ όλα μπερδεύονται. Υπάρχουν οι συνήθεις ένοπλες συγκρούσεις, υπάρχουν οι συγκρούσεις μεταξύ των γεωργών και άλλων ομάδων, των κτηνοτρόφων. Υπάρχει η λειψιδρία ούτως ή άλλως. Υπάρχει το κλίμα που πιέζει άπαντες και πιέζει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη γη τους. Υπάρχει εισαγωγή όπλων από τα υπολείμματα του Λιβικού στρατού. Το Μαλί δεν θα υφίστατο καν ως χώρα αν δεν είχε παρέμβει η Γαλλία. Ε, θα είχαν συμβεί αυτά που συνέβησαν με την Άισις στο Ιράκ. Και η Γαλλία είχε δίκαιο που ζητούσε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν σε μια παρέμβαση που δεν είναι μεταπικιοκρατική. Γιατί ακούμε και τέτοια. Και υπάρχει και ένα παρελθόν ιστορικό. Αλλά αυτά που συμβαίνουν εκεί είναι απειλή για μας. Δεν έχει καμία σχέση με το απικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας. Τα σύνορα της Ευρώπης είναι στο νότο της ε, Σαχάρα υπό την έννοια αυτή. Και θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Υπάρχουν κάποιες ομάδες ε, μη εμπόλεμες από τη Γερμανία, υπάρχουν κάποιοι άλλοι σύμβουλοι ε, Βρετανοί και Ισπανοί αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση στο Σαχέλ, θα, θα πρέπει να αναπτύξουμε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες η Γαλλία από μόνη της δεν δύναται να το κάνει. Θα έχουμε ομοφωνία για να προχωρήσουμε σε ειρηνευτική αποστολή ευρωπαϊκή. Δεν φοβούμε πως δεν νομίζω. Με κανόνα ομοφωνίας δεν πρόκειται να δούμε ευρωπαϊκή αποστολή τέτοια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως μια συμμαχία of the willing που λέμε αυτοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και βεβαίω οι λύσει δεν είναι μόνο στρατιωτικέ επιχειρήσει. Εκεί χρειάζεται υποστήριξη ε, για να δημιουργηθούν κρατικέ δομέ. Αλλά πώ να γίνει αυτό σε μια χώρα που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια σε κανέναν απολύτω. Εγώ πράγματι εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε λοιπόν και άλλες δυνάμεις και άλλες χώρες. Ουκρανία. Θα δούμε και με την ε, τετράδα της ε, Νορμανδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απουσιάζει. Γιατί ξέρετε υπάρχουν κάποια βήματα στα οποία απουσιάζουμε. Εν πάση τόσο η Γαλλία και η Γερμανία ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες. Το συζητήσαμε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας στο Τόκιο πριν από λίγες ημέρες. Όσο δηλαδή Υπουργό Εξωτερικών Τη ισπανία δεν ξέρω που θα οδηγηθούμε, αλλά είναι προφανές τουλάχιστον κατ' εμέ ότι με τη Ρωσία θα πρέπει και να διατηρήσουμε την πολιτική των κυρώσεων εφόσον δεν έχουμε πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα ε, να μην αγνοούμε, να μην αρνούμαστε την ύπαρξη μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία μας παρέχει και ενέργεια και με την οποία πρέπει να έχουμε σχέσεις. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα, συντεταγμένα και αυτό περνάει από την πλήρη υποστήριξη που πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία ώστε να ανθίσταται της πολεμικής πίεσης, της εισβολής και της ανάκτησης του ελέγχου στον Τονπάς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν είμαστε ενωμένοι, αν έχουμε ενωμένη θέση απέναντι στη Ρωσία. Και μέσω των πρωτοβουλίων της Γαλλίας ενισχύθηκε αυτή η ενοποιημένη θέση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε συσχετισμούς. Γιατί μπορεί κανείς να είναι και θαραλέος και φιλόδοξος και ευγενικό. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή γραμμή, μια σταθερή θέση, να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. προς την κυρία Βιγιανουέβα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να προσθέσω στα όσα ήδη είπα για την ε, Νότια Αμερική, γιατί εκεί υπάρχει πολύ σημαντική κοινωνική κρίση. Ε, και λέω ειλικρινώς ότι δεν γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια τι δυνατότητες θα είχε για να παρέμβει σε αυτή την κρίση που εξεράγει με τρόπο απρόβλεπτο, λέει ο κύριος Μπορέλ, το πιο επίγον κατά την άποψή μου είναι το θέμα της Βενεζουέλα. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο προδραστικοί. Γιατί το 1 τρίτο του πληθυσμού ε, αντιμετωπίζει το φάσμα της ασυντίας Το οποίο είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κυρώσεων που επηρεάζει τον πληθυσμό της χώρας. Που εμείς δεν το έχουμε εφαρμόσει, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείες ναι. Έχουμε οδηγηθεί σε ένα διέξοδο όπου αυτοί που πληρώνουν που πληρώνουν την ύφη είναι οι κάτοικοι της χώρας. Προφανώς δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα για, το, για την πολυμέρεια, γιατί δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι απλώς ρητορικά μιλώ. Δεν υπάρχει εναλλακτική στο σύστημα της πολυμέρειας και οπωσδήποτε η απάντηση, η εναλλακτική λύση στην πολυμέρεια δεν είναι η μονομέρεια. Γιατί αυτό απλώς σημαίνει ότι είναι ότι περνάει ο κανόνας του ισχυρότερου. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε το κράτος δικαίου, θέλουμε νόμους, θέλουμε μια δίκαιη προσέγγιση προς την προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων στα διάφορα μέρη του κόσμου και στην Νότια Αμερική όπου υπάρχει, ξαναλέω, οξύτατη κρίση κοινωνική. Και αυτά τα προβλήματα μπορεί να τα λύσει μόνο η δημοκρατία και τίποτε άλλο. Τώρα θα πολύ θα χαιρόμουν να συνεχίσω να συζητώ μαζί σας, αλλά με περιμένουν στην Μπρατισλάβα και θα πρέπει να αποχωρήσω φοβούμαι. Λέει ο Μπορέλ. Κύριε Μπορέλ, λέει ο πρόεδρος, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αναχωρήσετε. Μας είχαν υποσχεθεί από το γραφείο σας 10 λεπτά ακόμα. Εγώ είμαι στις διαταγές του γραφείου μου και επομένω θα κάνω αυτό που σα είπε το γραφείο μου. Αν είπαν αυτό, τότε είχαν δίκιο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κόουλς από την Λετωνία παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ απλό το ερώτημά μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο είναι και αυτή που είπε περισσότερο υποστηρίζει τα ανθρωπιμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το διεθνής κτλ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη του είπα του εκπροσώπου ό,τι αφορά την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού νόμου Μαγνίτσκι. Ποια είναι η άποψή σας, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, θα διεύρυνε την εργαλειοθήκη ε, του 21ου αιώνα για να αντιμετωπιστούν ε, αυτά τα προβλήματα των κατάφορων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ε, πλέον τον ε, κύρο στη Ρωσία για παράδειγμα για διάφορες παραβιάσεις αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί η θέση σας ως έπατε που έχει να κάνει ακριβώς και με την επιβολή κυρώσεων και τον εντοπισμό αυτών οι οποίοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια είναι η αποψή σας για την οθέτηση ενός ευρωπαϊκού του νόμου Μαγνίτσκε Και το δεύτερο, πιο πολύ ε, είναι μια πρόσκληση προς εσάς ε, να σπάσετε την αρνητική πρακτική ε, της προκατόχου σας και να έρχεστε να έρθετε στο, στην ΚΕΠΑΠ της 2 στις 4 Μαρτίου ε, στην Κροατία. Να είστε εκεί αυτοπροσώπος ε, γιατί στο CFSP συγκεκριμένα είναι σημαντικό να έρθετε γιατί ε, πρέπει να ανταλλάσσετε απόψεις και με τα εθνικά κοινοβούλια. Ήταν αρνητική η πρακτική προκατόψης, ελπίζω εσείς να την εγκαταλείψετε. Επόμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φάμπιο Καστάλντο. Thank you, Chair. Estimado Alto Representante, querido Josep. Αγαπητέ κύριε Μπορέλ, πολύ χαίρομαι συγχαρητήριά μου, τα σερμά μου συγχαρητήρια για την ανάλυση των καθηκόντων σας ε, και επιτρέψτε μου να συνεχίσω τώρα στη μητρική μου στα Ιταλικά. Έχουμε λοιπόν μια κοινή θέση από το 2008 ο ύπατος εκπρόσωπος όμως ε, δεν κατάφερε να πείσει τα κράτη-μέλη να πείσουν, να τηρήσουν τα κριτήρια αυτά και γι' αυτό έχουμε την έλλειψη μηχανισμού κυρώσεων για τις χώρες εκείνες που δεν συμμορφώνονται. Εσείς ε, θεωρείτε ότι αυτή η θέση δεν πρέπει να επικαιροποιηθεί και με τις νέες τεχνολογίες, ε, την τεχνητή νοημοσύνη, τον κυβερνοχώρο, τα φωνικά όπλα τα νέας γενιάς που έχουμε δεν θα πρέπει να έχουμε αναλογικά μέτρα προληπτικά για χώρες που δεν τηρούν αυτήν την κοινή γραμμή. Επίσης θα ήθελα μία σκέψη από πλευρά σας για την Τινησία που ήμουν και επικεφαλής ε, αποστολής παρατήρησης ε, πρόσφατα ε, ώστε να είναι η παρουσία μας εκεί πιο ισχυρή στην άμεση μεσογειακή γειτονία. Εταιρική σχέση που είναι από τις πιο σημαντικές, τουλάχιστον υπό τη δημοκρατική έννοια στην άμεσο νότο μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Φον Χάλφορτ από τις κάτω χώρε. Δείξτε μας ε, έτσι και που είστε ακριβώς. Κουνήστε λίγο το χέρι να σας δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Κίνα, διότι σήμερα στι Ολλανδικές εφημερίδες ε, γράφει ότι σε ένα νοσοκομείο στο Ρότερνταμ ένας Κινέζος ερευνητή. Ε, που εργάζεται και στο Ροτενταμ και Πεκίνο ε, εργάζεται και το έργο του θα χρησιμοποιηθεί από Κινέζους που θα μπορούν να εντοπίζουν ε, τους Ουιγούρους και τους αντιφρονούντες με το έργο του. Ισχύει αυτό. Και αν είναι, βλέπουμε πώς σκέφτεται η Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για την εθνική κυριαρχία και ακαιρεότητα ή την αμοιβαιότητα στις διμερείς σχέσεις. Αν λοιπόν συνομιλούμε με την Κίνα ή με τον Κινέζο πρέσβη και αναφέρουμε το θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική οπτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν νομίζω και αυτοί υπογράψει την Οικουμενική Δεξιά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα αυτό είναι μια κοινή βάση συνεννόηση. Ε, τώρα, είπα, λένε ότι λόγω των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη μεταχείριση των Ουιγούρων ε, θα επιβάλλουν κυρώσει ε, στην χώρα αυτή. Εσείς τι θα κάνετε. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Μπορέλ. Κίνα, την Ισία, ό,τι θέλετε. Διαλέξτε και πάρτε. Ο Μπορέλ, κυρώσεις ε, είναι κάτι δύσκολο διαχειρίσιμο, ε, πάντοτε. Έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, με την επιβολή ρώσεων το παράδειγμα της Βενεζουέλας θα σας δώσω. Οι κυρώσεις που συλλογικά πλήττουν ένα λαό, δεν είναι και τόσο βέβαιον ότι θα φέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και προκαλείται οδύνη και πόνος στη χώρα. Τώρα, κυρώσει κατά συγκεκριμένων προσώπων είναι κάτι το οποίο εμεί κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επιβάλει πολλέ τέτοιε κυρώσει και από ό,τι κατάλαβα εσείς λέτε αν υπάρχει ε, ενδεχόμενο να επιληθούν κυρώσεις ε, σε αυτούς οι οποίοι ε, έχουν προβεί σε παραβάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα και τη Ρωσία. Εγώ θέλω συγκεκριμένα, συγκεκριμένες περιπτώσεις και υποθέσεις να μας φέρετε. Δεν μπορώ να δώσω μια γενική απάντηση. Σίγουρα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των συνομιλών μας με την Κίνα. Είμαστε προσελωμένοι σε αυτό και πρέπει να σας πω ότι ε, εντάξει, οι Κινέζοι μπορεί να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, είπατε όμως και εσείς ότι έχουν προσογράψει σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ακριβώς πάνω σε αυτό βασίζονται και οι συνομιλίες μας, οι συνομιλίες μας για αυτά τα θέματα. Προς το παρόν δεν είναι επιτάπητος στο Συμβούλιο ή πρόταση επιβολής κυρώσεων για τον τρόπο, ε, με τον τρόπο που εσείς ε, υπονοείτε τουλάχιστον. Τώρα το Μαγνίτς και αυτό που είπατε δεν το ξέρω ακριβώς αυτό το νόμο που λέτε. Νόμος Μαγνίτσκι. Έχει χάσει τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, έχει πεθάνει, τι είναι. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω περί πρόκειται. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε. The one who put the question Αυτός που έθεσε το ερώτημα μπορεί να το επαναλάβει. Κύριε Κόλτς, εσείς ε, για το νόμο Μαγνίτσκι που ρωτήσατε, μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημά σας. Ναι, βεβαίως. Ο νόμος Μαγνίτσκι λέγεται έτσι δηλαδή. Είναι ένα εργαλείο που έχουν κρίνει κάποιες χώρες για να εντοπίζουν παραβάτες των δικαιωμάτων και να τους ε, ζητούν να λογοδοτήσουν ενώπιν της δικαιοσύνης με άλλα μέτρα. Νομίζω ότι εν μέρει εφαρμόζεται αυτό ο νόμο ε, σε ΙΠΑ, Καναδά ε, και κάποια κράτη-μέλη της Ευρώπης, έξι συνολικά νομίζω. Υπάρχει μια ιδέα, ένα παρόμοιο εργαλείο να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το ερώτημα είναι αν εσείς θα υποστηρίζετε μια τέτοια πρωτοβουλία εφόσον ε, ε ο εκπρόσωπος πρέπει να παρακολουθεί και τι γίνεται στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και ποιες παραβιάσεις διαπιστώνονται. Ευχαριστώ κύριος Μπορέλ. Δεν έχω επαρκή ενημέρωση για το θέμα και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μου λέτε αν υποστηρίζω αυτή την ιδέα ή αν θα πρότεινα στο Συμβούλιο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν ένα τέτοιο νόμο που λέτε έξι ευρωπαϊκές έχουν πάρει μια τέτοια απόφαση μου. Όχι, κοιτάξτε, πρέπει να το μελετήσουμε πρώτα απαντήσουμε. Okay, colleague uh, uh, this, the Committee Σήμερα το πρωί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε την ειδήσια έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλεια τη Ένωση. Και εκεί έχουμε αναφερθεί ε, στην ε, εισαγωγή του νόμου Μακρίτς και είναι μια μακρά συζήτηση, ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών. Τα άλλα ερωτήματα για την Κίνα, για παράδειγμα. Δεν απάντησα, απάντησα κ. Μπορέλ. Κύριε Καστάλτο. Για την Τινησία εσείς είχατε ρωτήσει. Η Τινησία ήταν η επαρχή της Αραβικής Άνοιξης. Και είναι η μόνη χώρα που επέζησε μετά από αυτήν την Αραβική Άνοιξη και δεν ξανάπεσε σε δικτατορικό καθεστώς. Η Τινησία λοιπόν είναι μια μεγάλη ελπίδα για τη δημοκρατία στη Βόρεια Αφρική και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην σβήσει η φλόγα της δημοκρατίας στην Τινησία. Γνωρίζετε, είπατε καλά τη χώρα αυτή και εγώ τη γνωρίζω καλά και νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα φάρο ελπίδα για τη δημοκρατία στην Βορεια Αφρική. Και όπω σα είπα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, διατηρήσουμε την ελπίδα. Για ε, μια χώρα που καλύτερα από τις άλλες ε, ξεπέρασε την κατάσταση που πρόκειψε μετά από ε, τη δημοκρατική αυτή έκρηξη του 2011 που δυστυχώς άλλες χώρες ε, ε, δεν διατηρήθηκε. Έσβησε αυτή η φλόγα. Okay, thank you. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπορέλ. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση με του εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστούμε που τι απόψει και απαντήστε τι ερωτήσει. Θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Ναι. Δεν απάντησα στην ερώτηση αν θα μεταβώ στην Κροατία. Θα χαιρόμουν πολύ να πάω στην Κροατία. Έτσι λοιπόν ήδη αναλαμβάνω αυτή τη δέσμευση και θα μεταβώ. Κύριε Μπορέλ, ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε ζωντανά στο Ζάγκρεμπ. Και είναι σημαντική αυτή η δήλωσή σας στο τέλος και είναι πολύ σημαντικό και για τους Κροάτες. Λοιπόν, έρχεται και ο Επίτροπος Βαρχέλη, θα έρθετε εδώ σε τρία λεπτά. Σας παρακαλώ να σας ζητήσω να επικεντρωθείτε κυρίως σε θέματα που αφορούν τη γειτονία και τη διεύρυνση, γιατί αυτή είναι, αυτά είναι τα αρμόδια, συγγνώμη, για αυτά τα θέματα είναι αρμόδιος ο κύριος Βαρχέλη. So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. So we now move to... Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος ε, της ε, σημερινής ε, συνάντησης. Και αφού είχαμε την ανταλλαγή απόψεων με τον είπα εκπρόσωπο, τώρα είναι ικανοποίησή μου να καλωσορίσω τον κύριο Όλιβερ Βαρχέλη, τον νέο Επίτροπο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Colleagues. Συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βαρχέλη Απλώ να σα ενημερώσω, κύριε Επιτροπέ, ότι έχουμε εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου, τη Βασνία Ερτζεγοβίνη και του Μαυροβουνίου. Επικεντρώνεστε ε, βάσει και του φακέλου σα στην πολιτική διεύρυνση. Θα ήθελα να ενημερώσω αδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερου. Έχω ένα κατάλογο με ονόματα και προσπαθώ εδώ να τα ελέγξω φυσικά. Προτεραιότητα έχουν οι συνάδελφοί που έχουν ζητήσει το λόγο για τον πρώτο γύρο. Θα προσπαθήσω να είμαστε δυνατόν πιο δίκαιος και χωρίς χρονοτριβή. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Και όσο περισσότερο χρόνο δώσετε στους συναδέλφους για τη συζήτηση, τόσο πιο ικανοποιημένοι θα επιστρέψουν στις χώρες τους και θα μιλάνε θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου και να επικεντρωθώ στα απολύτως απαραίτητα. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, καλωσορίζω την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια, τόσο σύντομα αφού ανέλαβα καθήκοντα. Είναι μία από τις πρώτες ανταλλαγές απόψεων που έχω. Χθες είχα την ευκαιρία να συναντήσω τα μέλη των Κοινοβουλίων των Δυτικών Βλυκανίων σε αυτή την Επιτροπή και σήμερα είμαι ιδιαίτερα ε, χαρούμενος που συναντώ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ζωτικό ρόλο στην Ευρώπη στην πολιτική της διεύρυνσης. Η διεύρυνση δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς ε, τη συνένεση των Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτό το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη όταν ε, σχεδιάζω το έργο που έχουμε νοποιών μας. Χθες συζητήσαμε με τους συναδέλφους από τα Δυτικά Βαλκάνια το πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για αυτούς και για μας. Σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική και στο κοινό μας μέλλον. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές. Οι χώρες αυτές βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης. Το να υποστηρίξουμε την περιφέρεια είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Όλοι θα κερδίσουμε αν ευημερούν οι άμεσοι γειτονέ μας, αν είναι ασφαλεί και σταθεροί. Όλοι εποφελούμαστε αν η οικονομία στην περιοχή είναι ισχυρέ. και υπάρχει ευημερία και πριν την προσχώρηση. του ίδιο ισχύει για την διασυνδεσιμότητα σε τομέα μεταφορών, ενέργεια ή ψηφιακά. Επίσης, οι χώρε των Δυτικών Λοκανίων έχουν συνεργαστεί καλά για τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση μαζί μας, αλλά χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο μεταναστευτικό. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να δώσουν και πολύτιμες συμβουλές στα κοινοβούλια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μπορούν να τις βοηθήσουν να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, να προωθήσουν την κοινοβουλευτική λογοδοσία, την εποπτεία του εκτελεστικού σώματος και τον δημοκρατικό έλεγχο. Ο καλύτερος ε, τρόπος να προωθήσουμε την πρόοδο στην περιοχή που αποτελεί ε, μέρος της Ευρώπης είναι μέσω μιας αξιόπιστης διαδικασίας διεύρυνσης. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η προοπτική προσχώρησης παραμένει αξιόπιστη. Καταρχήν, οι μεταρρυθμίσεις που ε, υλοποιούν όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να έχουν πραγματικό αντίκτυπο επιτόπου. Αυτό σημαίνει δηλαδή να υπάρξει ευμερία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και το αίσθημα της ελευθερίας στις χώρες εταίρους. Αυτό θα συμβεί μόνο αν ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων ε, ε όχι απλώς διατηρηθεί, αλλά επιταχυνθεί. Αξιότιμα μέλη, νωρίς ε, του χρόνου η Κομισιόν θα προετοιμάσει προτάσεις για να συνεισφέρει στο να προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία και να βασιστεί στην περσινή στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, να ενδυναμωθεί η συνεργασία και η διαδικασία διαπραγματεύσεων να γίνει πιο αποτελεσματική ενώ ταυτόχρονα θα απαντήσουμε και στις ανησυχίες κάποιων κρατών μελών. Λοιπόν, ε, τα θεμελιώδη στοιχεία του κράτου δικαίου, οικονομική ανάπτυξη, λειτουργία δημοκρατικών θεσμών ε, και μεταρρύθμιση τη δημόσια διοίκηση ε, θα βρίσκονται ψηλά στην ημερησία διάταξη. Αυτά είναι θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης της κοινωνίας που υφίσταται όλε οι κοινωνίε των Δυτικών Βαλκανίων για να είναι έτοιμε για την προσχώρηση. Πέρα από την εστίαση σε αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, θέλω να είναι πιο δυναμική η διαδικασία και όχι απλώ να επικεντρώνεται στην έναρξη στο κλείσιμο κεφαλαίων. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες ε, για ε, πιο στενή και νωρίτερη ολοκλήρωση. Τα κίνητρα είναι απαραίτητα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θέλω να δω να ενταχθεί καλύτερα η περιοχή σε βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και πριν την ένταξη. Παραδείγματο χάρη, τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να σχετίσονται στενά με τον Green Deal, με το ψηφιακό θεματολόγιο ή με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στην ενέργεια και στις μεταφορές. Οι λαοί της περιοχής δεν θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την προσχώρηση για να δράξουν το ωφέλη αυτών των βασικών πολιτικών η πολιτική δέσμευση χρειάζεται για τις μεταρρυθμίσεις στην περιοχή, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να δω καλύτερη διαχείριση της πολιτικής διαδικασίας και στενότερη συμμετοχή των κρατών μελών, ακόμη και σε υψηλότερο επίπεδο, για να υποστηρίξουμε τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται οι κυβερνήσει ε, στην περιοχή θα πρέπει να αναλάβουν ε, την ευθύνη έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι συμμετοχική η διαδικασία. Τα κοινοβούλια έχουν ρόλο κλειδί σε αυτή τη διαδικασία, όχι απλώ να μπορούν ε, να ελέγχουν τι κύριε νομοθετικέ προτάσει μεταρρύθμιση που θα παρουσιάζονται ενώπιόν του. και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχτεί νέα μέλη όταν πληρούνται οι προποθέσει. Αυτό δεν θα πρέπει να επιβραδύνει τη διαδικασία τη προσχώρηση κατά κανένα τρόπο. Οι δύο διαδικασίες που δίνουν η εμβάθυνση δηλαδή της ολοκλήρωσης και η προσχώρηση μπορούν να τρέχουν παράλληλα. Περιφερειακή συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονία είναι ζωτικές για την πρόοδο των χωρών στην Ευρωπαϊκή Οδό. Εγώ στο πλαίσιο αυτό θα υποστηρίξω πλήρως την επίλυση διμερών διαφορών. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τον είπατο εκπρόσωπο, τον Ιωσεπ Πορέλ, με το στόχο να επαναφέρουμε το διάλογο Πριστίνας Φελιγραδίου σε μια επιτυχία εκβασίδη του χρόνου. Αξιότιμα μέλη, πρόσφατη έλλειψη συνένεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις προσχώρηση με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ήταν πηγή απογοήτευση για πολλού από εμά. Παρ' όλα αυτά, η δέσμευσή μα στην ευρωπαϊκή του προοπτική παραμένει μετάβλητη. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστα γεωπολιτικά ω Κομισιόν αν ε, δεν διορθώσουμε τι σχέσει με τους άμεσου γείτονε μα. Και τα Δυτικά Βαλκάνια είναι κάτι παραπάνω από γείτονε, βρίσκονται στην καρδιά τη Ευρώπη. Θα συνεχίσω να υπερασπίσω την πρότασή μας να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης και με τις δύο χώρες και δεν μπορώ παρά ε, να τονίσω τη σημασία της θετικής απόφασης να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, στην Σύνοδο του Ζάγκρεπ του χρόνου. Η Προεδρία της Κροατίας λοιπόν θα έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω και δύο λόγια για την Αλβανία και την υποστήριξή μας στη χώρα κατόπιν του σεισμού της περασμένη εβδομάδας. Αμέσως ξεκινήσαμε ε, να ενεργοποιούμε το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας ε, και πολλά κράτη-μέλη έδωσαν βοήθεια επί τόπου μετά την καταστροφή. Επίσης, εξετάζουμε πώς θα βοηθήσουμε πέρα από την κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση του Σώματος, αποφασίσαμε να δώσουμε 50 εκατομμύρια ευρώ στην Αλβανία ως ε, βοήθεια ε, μετά την καταστροφή και θα οργανώσουμε και μια σύνοδο δωρητών για τη χώρα και εξετάζουμε και περαιτέρω δυνατότητες να βοηθήσουμε την Αλβανία για να ε, ανακάμψει από αυτή την καταστροφή. Πρόεδρε, να κλείσω με ένα σχόλιο για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή η Επιτροπή ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των πολλών αλλαγών, των οποίων θα γίνουμε μάρτυρε, ε, καμία δεν θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από ότι το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Πιστεύω ενθερμά ότι ο συνδυασμό ε, τη νέα Επιτροπή και του νέου πολιτέ δημοσιονομικού πλαισίου θα φέρει ανανεωμένε ευκαιρίε για στενότερη συνεργασία με του εταίρου μα και επίσης θα αυξήσει την δυνατότητα επιρροής μας ε, στην περιοχή. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Thank you, Oliver Um, the format is here I give the floor and as many colleagues as possible can... Προσπαθήσω να δώσω ε, το λόγο σε όσο το δυνατόν στους συναδέλφους εσείς θα μας πείτε πότε θέλετε να σταματήσουμε για να απαντήσετε και να συνεχίσουμε τους επόμενους γύρους από τα Εθνικά Κοινοβούλια Φασίνα που είναι ο πρώτο ομιλητής. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Εκτιμώ τα όσα είπε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Επίτροπος πρέπει να έχουμε συνείδηση του εξής. 24 ε, χρόνια πέρασαν από την Συμφωνία Ειρήνευσης του Ντέιτον, την επόμενη μέρα της οποίας εμείς είχαμε υποσχεθεί, εδώ είμαι, Επίτροπε, ε, είχαμε υποσχεθεί, λέω, στις χώρες εκείνες, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προϋπόθεση η ειρήνευση και η σταθερότητα στην περιοχή. 24 χρόνια είναι ένα τέρτο του αιώνα. Έχουν γεννηθεί δύο γενναίες. Εάν εμείς αναβάλλουμε και αναβάλλουμε και αναβάλλουμε, θα έχει απλώς την εξής επίπτωση. Θα υπάρξει αγανάκτηση, θα υπάρξει έλλειψη εμπιστοσύνης, θα μειωθεί το επίπεδο της φιλοδοξίας και της προθυμίας ένταξης και θα παραχωρήσει έδαφος στο λαϊκισμό. Ε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση του Επιτρόπου, δηλαδή και πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ, θα πρέπει να απομακρυνθεί η, θέση μπλοκ που αποφάσισε το Συμβούλιο για την Αλβανία και τη Βορρία Μακεδονία. Ε, ε, συνάδελφοι, διακόπτει ο Πρόεδρος, έχουμε κανόνες. Ναι, μιλούμε για τον Επίτροπο Διεύρυνσης και Γειτονικών Χωρών. Τι πιστεύετε για την κατάσταση στη Μεσόγειο και για το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γκάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε στην εισαγωγή σας παρέμβαση. Ξεκάθαρα είπατε ότι φυσικά θα πρέπει πρώτα να πληρούνται προϋποθέσεις και μετά να προσχωρήσει κάποιο και να κριθεί με βάση το τι έχει πετύχει για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία όμω γιατί θεωρούνται αυτές οι χώρες ως πακέτο και δεν κρίνεται με βάση ε, ε, το, το τι έχει πετύχει κάθε χώρα ξεχωριστά. Γιατί ξέρετε ότι ακούστηκε και κάποια κριτική σε ό,τι αφορά τι εξέλιξη στην Αλβανία. Ίσως και αυτό ήταν ένα από τους λόγους ε, που ο Γάλλος Πρόεδρος τελικά είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμονή. Μήπως θα πρέπει να ε, σπάσει αυτό το πακέτο για να δοθεί ένα πολιτικό μήνυμα. Ε, να ξεκινήσουμε ενδεχομένω με τη Βόρεια Μακεδονία, να μην χαθεί ο ρυθμός, η όθηση και έπειτα να προχωρήσουμε. Αυτό έγινε κατά το παρελθόν. Ε, είχαμε δύο γκρουπ, δύο ομάδες στις χώρες μέλη Κεντρικής Ευρώπης και μήπως θα μπορούσε να επαναληφθεί αυτό το μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχαήλ Γκάλε, ο πρόεδρος από τα Εθνικά Κοινοβούλια επόμενη συγκεκριμένη και ταγκούι από τη Γαλλία. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σχετικά με μια δήλωση που μόλις κάνατε, είπατε ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση μπορούν να προχωρήσουν παραλλήλως. Η Γαλλία, ωστόσο, μπλοκάρει το άνοιγμα διαπραγματεύσεων ένταξη, Παράλληλα έχει υποβάλει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε μια σταδιακή διαδικασία ένταξης ή προσέγγισης με συγκεκριμένα πρότυπα διακυβέρνησης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπη εν ώψη και τη συνόδου του Ζάγκρεπ, ε, πώς βλέπετε την γαλλική πρόταση. Θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες οι χώρες αυτές σε διαρθρωτικά κονδύλια. Και επίσης πώς βλέπετε και το ρόλο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πρόοδου των υποψηφίων χωρών. Αναφερθήκατε στον προϋπολογισμό του 2020 που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, που προβλέπει και ένα φάκελο για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αυτά τα πρόσθετα κονδύλια πώς θα κατανεμηθούν, Επίτροπε. Ε, ποιες θα είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες για καλύτερη συνεργασία και ένταξη των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία μου, λέει ο πρόεδρος. Σάντσε Σαμό για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε τον κύριο Μπορέλ προηγουμένως. Αναφέρθηκε στην Τουρκία σε τέσσερις περιπτώσεις. Ο κύριος ε, Βάρχελη ε, λέγει ότι ε, θα συνεργαστεί στενά με τον κύριο Μπορέλ για την Τουρκία. Αυτή η διπλή πταχή, η πτυχή με η διάσταση της Τουρκίας, γείτονα και σημαντική χώρα αλλά και υποψήφια, δεν ξέρω μήπως είναι μια διτή ταυτότητα τις οποίες πρέπει να συμφωνήσουμε, να συνοηθούμε καλύτερα, πώς θα κατανεμνύμετε μεταξύ σας τις αρμοδιότητες της προσέγγισης αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάρχελη ζήτησε ομάδες πέντε ερωτήσεων. Έχω λοιπόν και τον κύριο Πίσκο από την Πορτογαλία. Είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχα κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μπορέλ, δυστυχώς δεν πρόλαβα να το τις υποβάλω, αλλά και για τη μελλοντική διεύρυνση έχω κάτι ερωτήσεις. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν φρονιμότερο να δοθεί περισσότερο χρόνος στις υποψήφιες να ανακτήσουν έδαφος στο επίπεδο των ευρωπαϊκών εξιών προτού ενταχθούν. νομίζω ότι έχουμε αντιπροσωπείες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, θέλω να σας πω κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφο που είχαμε μόνο 20 λεπτά να υποβάλουμε ερωτήσει στον κύριο Μπορέλ. Την επόμενη φορά θα εκτιμούσα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Δεν είμαι υπεύθυνο για το χρόνο του είπα του εκπροσώπου. Αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που είχε ακόμα και χρόνο να έρθει μέχρι πριν από δύο εβδομάδες ε, δεν ήμασταν καν βέβαιοι ότι θα είχαμε νέα επιτροπή. Έτσι συνολικότερα. Ο κύριος Βάρχελη τελικώς ε, τα κατάφερε στο δεύτερο γύρο ε, και είναι ενδεικτικό αυτής της κατάστασης. Έχουμε πολλούς συναδέλφους κύριε Βάρχελη που θέλουν ακόμα το λόγο. Ε, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται στις απαντήσεις μου για να έχουμε το μέγιστο αριθμό ερωτήσεων από την αίθουσα. Για την ερώτηση του κυρίου Γκάλα, για την αποσύνδεση είναι ένα πολιτικό προϊόν θα έλεγα το οποίο βλέπουμε να ανέρχεται ή να κατέρχεται ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες, επιτρέψτε μου αυτήν την έκφραση. Πρέπει όμως να δούμε τις χώρες κάθε μία για την περίπτωση τη δική της, με τα υπέρ και τα κατά που έχει. Έχουμε ένα σύνολο προδιαγραφών και για τη Βόρειο Μακεδονία και για την Αλβανία, τις οποίες έχουν καλύψει. Επομένως το να συνδέονται ή όχι, το να γίνεται coupling ή όχι, έχουν καλύψει, έχουν συμμορφωθεί. Και γι' αυτό πρέπει από κοινού να λαμβάνουμε την απόφαση. Θα ήμασταν άδικοι προ τη μία ή την άλλη χώρα, εφόσον δεν επιβραβεύαμε τα ίδια επιτεύγματα με τον ίδιο τρόπο. Η προσέγγιση μου εξακολουθεί να είναι και θα εξακολουθήσει να είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε διαπραγματεύσει το Μάρτιο και με τις δύο αυτές χώρες. Βεβαίως, δεν έχω προβλήματα ακοής. Ακούω τι ανισχύσει που εκφράζονται από διάφορα κράτη-μέλη σχετικά με την Αλβανία και θα εξασφαλίσω ότι θα έχουμε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Δεν πρόκειται να τα καταφέρω θα προσεγγίσουμε τις χώρες αυτές και αν χρειαστεί και τα εθνικά τους κοινοβούλια. Ε, συναντήθηκα και με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Δανικού Κοινοβουλίου. Θα κοιτάξω να κάνω ό,τι γίνεται για να βρεθεί μια λύση. Για τη γαλλική πρόταση, να πω. Υπάρχουν και πολλές άλλες, έτσι, επιτάπητος, όχι μόνο η γαλλική υπάρχει και σημαντική ομάδα κρατών μελών που είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένα σχετικά με την έλλειψη απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά, όπως είπα, πρέπει να δούμε και τι ανησυχίε τους. Εγώ θα το κάνω, θα επισκεφθώ το Παρίσι πολύ σύντομα, θα μιλήσω με τους Γάλλους αρμοδίους για να καταλάβω τις ανησυχίε τους, αλλά και οι γαλλικέ αρχές είναι σαφεί ω προ το εξή. Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει την ενωσιακή προοπτική των χωρών αυτών. Αυτό δεν το θίγει κανείς. Δεν πρέπει να ανοίξουμε καμία συζήτηση λοιπόν και δεν πρόκειται να το κάνουμε ως προς αυτό. Μπορώ να δω τη μεθοδολογία, μπορώ να δω πώς καλύτερα μπορούμε να συσχετίσουμε την πρόοδο των χωρών αυτών με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις κυβερνήσεις, πώς μπορούμε να ομαδοποιήσουμε την προσπάθειά μας και την αξιολόγησή μας, αλλά δεν πρόκειται να πάω σε συζήτηση επί της ουσίας για την προοπτική των χωρών αυτών. Για τον προϋπολογισμό, την αύξηση του προϋπολογισμού. Μπορεί να μας χρησιμεύσουν τα κονδύλια αυτά ώστε να εντάξουμε το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων στο δίκτυο TNT, το οποίο είναι κρίσιμο για τη μεγέθυνση οποιαδήποτε οικονομία γιατί χωρίς υποδομές ενεργειακές και μεταφορών δεν γίνεται. για την κοινή μας ε, συνεργασία με τον ύπατο εκπρόσωπο για την Τουρκία. Είναι προφανές ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων δρά κολεγιακά. με τον κύριο Μπορέλ τις τρεις πρώτες μέρες των καθηκόντων μας, ε, νομίζω τον συνάντησα δέκα φορές, αν με τις καλά. Ε, επί της Τουρκίας, είναι απλώς η πολιτική γειτονία που διακυβεύεται εδώ. Αλλά η εξωτερική πολιτική ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά και λειτουργούμε ως ομάδα, σας βεβαιώ. Για την δε κατάσταση για τη Μεσόγειο. Εδώ θα μπορούσα να μιλάω για πολλά περισσότερα λεπτά από ό,τι έχω στη διάθεσή μου. Πρέπει να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη και σε αυτήν την περιοχή και για αυτούς που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας πρέπει να δημιουργήσουμε τις οικονομικές συνθήκες μιας σταθερής κοινωνίας και για αυτούς που είναι πρόθυμοι να συνεργαστεί μαζί μας και για θέματα πολύ σημαντικά για μας που είναι η μετανάστευση, θα έχουμε την πιο στενή συνεργασία που μπορούμε. Για παράδειγμα, το Μαρόκο θα μπορούσε να είναι πρότυπο παράδειγμα για όλη την περιοχή. Θα είμαστε απολύτως ανοιχτοί να έχουμε αντίστοιχη, αντίστοιχα υψηλού επίπεδου συνεργασία και με άλλες χώρες, π.χ. την Τινησία. Θα Κάνουμε λοιπόν μια προσέγγιση, θα κάνουμε reaching out για να το πούμε ελληνικότερα, για να βρούμε και τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δεύτερος γύρος. Οι φίλοι από το Εθνικό Κοινοβούλιο έχουν το λόγο και πάλι. Πρώτος από την Πολωνία ο κύριος Κλίχ ή Κλίτς. Κλίστ. He's not here. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Αζουμπάλης από τη Λιθουανία. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ένα ερώτημα για την ενδεχόμενη κοινή θέση για να αποφύγουμε πλέον τις ε, μόνιμες προσπάθειες ε, της Ρωσίας να, να κόψει το δρόμο ορισμένων χωρών ε, στη, προς την Ένωση και δεύτερο για την ε, Λευκορωσία. Ξανά ασχολούμαστε με τη χώρα αυτή. Μήπως βοηθάμε την επιβίωση της δικτατορίας Λουκασέγκο. Ευχαριστώ. Κούτσο και ο Στρεβίτσιος. Ένας από τους δύο παρακαλώ, συμφωνήστε μεταξύ σας. Ο Πέτρας ή ο Έλαν. Να αντιμοιραστούμε την ερώτηση. Εντάξει, να αντιμοιραστεί 30 δευτερόλεπτα ο καθένας τότε. Ωραία, ωραία. Είμαστε στην ίδια ομάδα, το Renew. Και μπορούμε να ανανεώσουμε, όπως είμαστε του Renew, πολλά. Λοιπόν, μέχρι τα Χριστούγεννα, κύριε Επίτροπε, ίσως να έχουμε μια χώρα λιγότερη στην Ευρώπη. Μπορεί να την καταπιούν τη Λευκορωσία οι Ρώσοι. Κάθε μέρα συνεδριάζουν. Εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε γενικά ζητήματα. Ε, και εκεί γίνεται λόγος για ένταξη της Λευκορωσίας ε, στην Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, όμως εγώ θα το έλεγα τελείως διαφορετικά προσάρτηση ε, μιας χώρας ε, στον 21ο αιώνα. Ποιες είναι οι ε, επιπτώσεις από την εξαφάνιση μιας δημοκρατικής χώρας λοιπόν. Έλα, 30 δεύτερα, ε, Μ, ναι, το πετύχατε τώρα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτή τη γαλλική πρόταση, το non-paper, το ανεπίσημο αυτό έγγραφο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τι είπατε για τη μεθοδολογία και το πραγματικό ε, ουσιαστικά ερώτημα. Αν προτίθεστε να αλλάξει αυτή η μεθοδολογία, αν η απάντηση σα είναι θετική, είναι ναι, τότε σε επίπεδο επιτροπή Πώ αυτό μπορεί να γίνει και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ποια θα είναι η μελλοντική διευθέτηση, τι συμφωνία υπάρχει, πώς διαμορφώνται οι απόψεις. Και τώρα μία από τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν από το Μαυροβούνιο, Ρακολόσεβιτς. Πού είναι το Μαυροβούνιο? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Αυσπέσα να είμαι σύντομο. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εκπληρώσουμε όλες μας τις ε, και δεν θα καταλήψουμε το μέλλον μας. Ε, τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να είναι στην Ένωση. Βοηθήστε μας όμως ε, για να μην χάσουν ενθουσιασμό τους ε, οι κοινωνίες των χώρων των Δυτικών Βαλκανίων. Αν γίνει αυτό θα ανοίξει ο δρόμο σε τρίτες χώρες που έχουν τα δικά τους συμφέροντα και θέλουν να ασκήσουν επιρροή στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε πολύ καλά στο Μαυροβούνιο γιατί είχαμε τη ρωσική επιρροή τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημά μου το εξή. Γίνεται λόγος για μεθοδολογία. Αυτό τι σημαίνει. Θα αλλάξει η μεθοδολογία για τις χώρες που έχουν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία εδώ και 7 χρόνια διαπραγματευόμαστε εμείς στο Μαυροβούνιο ε, ήδη. Θα αλλάξει ή θα μείνει η ίδια η μεθοδολογία για τις χώρες αυτές που έχουμε ήδη ξεκινήσει ή δεν το γνωρίζετε ακόμα. Βέβαια, για όσε χώρε ξεκινούν τώρα ή μετά τι διαπραγματεύσει, φαντάζομαι θα ισχύει η νέα μεθοδολογία. Γιατί γίνεται για αυτέ που έχουν ήδη ξεκινήσει. Με Γουόλε, εξακολουθεί να είναι εδώ. Όχι, επόμενο. Μη γεγραμμένο. Γκέγκε ή κάπω έτσι από την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ για αυτή την uh, δυνατότητα που μας δίνετε να συνομιλήσουμε. Όπως αναφέρατε, η διαδικασία της διεύρυνσης ε, έλαβε ένα πλήγμα πριν λίγες εβδομάδες και μετά από αυτό το βέτο αναγνωρίσαμε ότι στα Βαλκάνια και στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το software ασκείται από πάρα πολλές χώρες ε, για να εκφράσουν την επιρροή τους ανάλογα με τη σφαίρα των συμφερόντων τους. Και να αναρωτιέμαι, ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία ασκούν τη δική τους επιρροή μέσω από πολιτιστικά ή οικονομικά μέσα και από πολύ συγκεκριμένε ιδέες και έργα. Τι έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από πολιτικά σλόγγαν στις χώρες που περιμένουν ε, την προσχώρηση. Δεύτερον, πόσο μπορεί να διατηρήσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία της διεύρυνσης, ενώ ζητά το σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων και ταυτόχρονα κάποια δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, ούτε σέβονται αυτές τις αρχές. Τρίτον, όταν εξετάζουμε τα μέσα που έχετε ως Επίτροπος στο να προωθήσετε περαιτέρω τη διαδικασία της διεύρυνσης, ποια είναι αυτά τα μέσα που έχετε για τους ε, μελλοντικούς υποψηφίους ε, αλλά και σε σχέση με τα κράτη-μέλη για να προωθήσετε το σεβασμό, στο, το σεβασμό των Να Ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και στην Ουκρανία αλλά και ε, στα κράτη της Βαλτικής και στα Βαλκάνια. Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριο Κουτσούμπας από την Ελλάδα στο 180, αν κάθεστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή, την πρόσκληση και να μεταφέρω εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Η πάγια θέση της ε, Ελλάδος είναι ότι υποστηρίζει την ενταξιακή προοπτική του συνόλου των χαρών των Δυτικών Βαλκανίων και της ευρύτερη περιοχή με σκοπό την διαφύλαξη της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Προϋπόθεση όμω για την εν λόγω ελληνική υποστήριξη αποτελεί η τήρηση αυστηρή αιρεσιμότητα βάσει των ιδίων επιδόσεων των υποψηφίων χωρών τη περιοχή. Θα ήθελα να κλείσω με έναν προβληματισμό. Μήπω όμω η διεύρυνση ή η συνεχεια συνέχιση ενταξιακών διαπραγματεύσεων των υποένταξη χωρών θα πρέπει να έχει ω προποθεση η προτεραιότητα την τήρηση του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα από, τα υποένταξη, από τις υποένταξη χώρες γιατί βρισκόμαστε τελευταία σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Second round. Ας περάσουμε στο δεύτερο γύρο, Όλιβερ. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ανατολική εταιρική σχέση. Προσπαθώ να μου ειδοποιήσω τις ε, ερωτήσεις για την Ουκρανία καταρχήν και για το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη συνεργασία και τη σταθερότητα με την Ουκρανία. Και πάλι πιστεύω ότι πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει φυσικά να υπερασπίζουμε την αδερφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας ε, και όσο δεν υπάρχει πρόοδος ε, στη διαδικασία του Μίνσκ δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τις κυρώσεις που έχουμε επιβάλει στη Ρωσία. Θα πρέπει επίσης ε, να δεσμευτούμε περισσότερο και να είμαστε πιο παρόντες στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, σε που θα ήθελε να συνεργαστεί βαθύτερα μαζί μας όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Φυσικά, όσες χώρες έχουν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, βαθιά και ολοκληρωμένη συμφωνία, μπορούν να εμβαθύνουν τις σχέσεις και είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό όμως ε, θα θέλαμε να ε, απευθυνθούμε περαιτέρω σε αυτές για την οικοδόμηση μιας οικονομίας της αγοράς. Και επαναλαμβάνω τα ίδια μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε και στα Δυτικά Βαλκάνια, ότι χωρίς πραγματική οικονομία οι χώρες αυτές πάντοτε θα είναι ευάλωτες και είναι προς το βέλτιστο συμφέρον μας να βελτιώσουμε τη σταθερότητα της περιοχής μας, της περιφερειάς μας, μέσω βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα, για τη Λευκορωσία. Η προσέγγιση μας είναι ότι όταν φύγουμε από οποιαδήποτε συνεργασία με τη Λευκορωσία θα χάσουμε και οποιαδήποτε επιρροή έχουμε. Ήδη έχουμε πολύ μικρή επιρροή στη Λευκορωσία Ήδη έχουμε έναν αυξανόμενο σωρευτικό ρυθμό συνεργασία μαζί του, αλλά πρέπει να είμαστε και επιτόπου. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε τι δικέ μα αξίε, γιατί διαφορετικά θα είμαστε κι εμείς ε, αυτοί που τελικά θα δεκτούμε τη στροφή τη χώρα αυτής προ τη Ρωσία. Όταν λοιπόν προσεγγίζουμε τη Λευκορωσία θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Για το γαλλικό έγγραφο, από ό,τι φαίνεται είναι σημείο αναφοράς για πολλού από εσά. Λοιπόν, η αλλαγή της μεθοδολογίας είναι το ένα. Τώρα το να αμφισβητεί κανείς όλη τη διαδικασία της διεύρυνσης είναι κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές στη μεθοδολογία για να είναι πιο αξιόπιστη και ε, για τις χώρες, ε, τις προσχώρες, αλλά και για τα δικά μας κράτη-μέλη. Αλλά αν το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είναι και πιο δυναμική η διαδικασία. Η δική μου λοιπόν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε αναθεώρηση της μεθοδολογίας θα είναι ότι όταν ε, οι χώρες ε, παρουσιάζουν αποτελέσματα και εμείς θα πρέπει να παρουσιάσουμε αποτελέσματα και είναι αυτονόητο γιατί είναι και μέρος της σημερινής μεθοδολογίας ότι αν έχουμε υπαναχώρηση τότε θα πρέπει και εμείς ε, να υπαναχωρήσουμε στις διαπραγματεύσει. Όμως δεν πρόκειται μόνο για το έγγραφο της Γαλλίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε και άλλες ιδέες. Τώρα, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις ε, για την διπλωματία, για το soft power και πώς ε, θα αυξήσει την επιρροή της η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Ακριβώς ε, γι' αυτό ανέφερα το οικονομικό επιχείρημα. Αν δείτε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Εμείς είμαστε μεγαλύτεροι επενδυτές στην περιοχή. Ε, δέχονται οι χώρες ε, αυτές ε, η επιρροή μπορεί να υπάρχει ένας συνδρομικός στάσιο, μια συνδρομική γραμμή ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, αλλά να έχουμε αυξανόμενη συμμετοχή στην περιοχή και μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για τις υποδομές, της μεταφορές, τότε θα έχουμε επιρροή στις χώρες αυτές τότε θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε αθέμητη επιρροή από τρίτες χώρες. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση, μεγαλύτερη επιρροή, αν ε, συμμετάχουμε περισσότερο. Αυτό είναι το σχέδιο που σας παρουσιάζω. Γιατί είναι αναθεώρηση της μεθοδολογίας. Έλαβα και μια ερώτηση αν το αν θα ίσχυε στις ήδη υφιστάμενες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση. Δεν νομίζω ότι είναι, ε, ότι είναι σοφή μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να αλλάξουμε τους κανόνες. Ποτέ δεν το κάνουμε, αλλά δεν θα ήθελα να το κάνω ούτε αυτή τη φορά. Φυσικά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δει το Σώμα των Επιτρόπων. Σχεδιάζουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη περιγραφή των ιδεών μας τον Ιανουάριο. Είναι υποσχεδιασμό αυτό και θα επανέλθω στην Επιτροπή σας ε, στη συνέχεια. Όμως σας διαβεβαιώ, δεν θα ήθελα να υπάρξει περαιτέρω επιβράδυνση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προωθήσω τη διεύνηση και να παρουσιάσω αποτελέσματα. Και τέλος, για τα συλλογικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, ναι, τα συλλογικά δικαιώματα για τις μειονότητες. Αυτά κάθε αυτά είναι ένα ζήτημα, δεν τα αναγνωρίζουν όλοι ως συλλογικά δικαιώματα. Είναι θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη τα δικαιώματα των μειονοτήτων ως συλλογικά. Παρόλα αυτά, η προστασία των μειονοτήτων είναι αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι εδώ για να την πίσω να την υπερασπίσω σε σχέση με οποιαδήποτε γειτονική χώρα και στα πλαίσια της διαδικασία της ε, διεύνησης. Αν δούμε την μειονότητα των Ρωμά στα Βαλκάνια, ως παράδειγμα, είναι ένα βασικό θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Η Ρωμά είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ιδιαίτερη μειονότητα στην περιοχή αυτή, με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Ναι, λοιπόν, ε, κύριε Γκέγκεσί, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, γιατί διαφορετικά η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και η ειρήνη θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτος γύρος. Πρώτος ομιλητής από τα Εθνικά Κοινοβούλια, Κάλνιντς από την Λετωνία. Yes, hello. Um, thank you very much. Um, Γεια σας, ευχαριστώ. Έχουμε μιλήσει για έναν αριθμό χωρών που είναι μέσα στην Ανατολική Γειτονία, αλλά για τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία δεν έχει ακουστεί κάτι. Έχουν κάτι κοινό δεν έχουν τελέσει κράτη μέλη της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχουν και τρεις κατεχόμενα εδάφη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το θεωρείτε φραγμό ε, στη μελλοντική τους ε, ενδεχομένως προσχώρηση στην ενωσή, τη σύνδεσή τους. Ξέρω ότι πρέπει να φέρουν σε πέρας κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα και θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη Γεωργία. Είναι μια χώρα που νομίζω θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Επαλεύει ακόμη. Ε, πρέπει να ε, τις αναγνωριστούν τα όσα έχει επιτύχει ήδη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βλάντιμιρ Μπουλτσικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που σας ε, βλέπω, κύριε Επιτροπέ, κάθε επιτυχία. Τρίτη μέρα πιάστε δουλειά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Κάποια σημαντικά για τη διεύρυνση ακούστηκαν και εσείς ξεκινήσατε την ομιλία σας ε, αναφερόμενη στα εθνικά κοινοβούλια και τα κοινοβούλια εν και το ρόλο τους και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Τι γίνεται όμως με τα Εθνικά Κοινοβούλια στα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ είμαι εισηγητής ε, για τη Σερβία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχω ε, με το, στο διακοινοβουλευτικό διάλογο. Όμως υπάρχει κατάσταση κρίσης στις χώρες σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, τη δημοκρατική κοινοβουλευτική παιδεία. Ποια είναι τα σχέδιά σα για να βοηθήσετε να βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα στεναρό πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για μεμονωμένε επισκέψει κτλ. Μιλάμε για το κράτο δικαίου. Ε, τα χρειαζόμαστε τα εθνικά ε, κοινόβουλια. Δεύτερον, να ε, μιλήσετε για τα οικονομικά ζητήματα. Όταν όμως βλέπουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την περιοχή, πολλές φορές είναι επιλεκτική και πιο πολύ γίνεται λόγος για το ρόλο της Ρωσίας και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Για την επικοινωνία λοιπόν, τι μπορεί να αλλάξει εν γέννη και πώς θα συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς των χωρών της περιοχής στην επικοινωνία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Επόμενος προσκεκλημένο από το Εθνικό Κοινοβούλιο, η κυρία Καρίμη από τις κατοχώρες. Oh, Πού είστε? Εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τι πληροφορίε που μα δώσατε και το ερώτημά μου έχει να κάνει με την Τουρκία. Δώστε μας λίγα παραπάνω στοιχεία γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια στεγανοποιημένη προσέγγιση απέναντι στην Τουρκία πρώτα σε ό,τι αφορά ε, τη μετανάστευση, το άσυλο μετά για την προσχώρηση στην ένταξη τρίτων για το ΝΑΤΟ. Σε διαφορετικά σιλό. Ε, γιατί και δεν έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Κύριε Επίτροπε, εδώ. I would rather use my mother tongue. μου Ερώτηση που υπέβαλε η συνάδελφός μου από το Λίβανο. Δηλαδή θα επικεντρωθώ στην Τουρκία. Το παράξενο με την Τουρκία είναι ότι δεν σέβεται ούτε καν τα θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Τουρκίας, δεν σέβεται το διεθνή δίκαιο και φυσικά δεν σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, του ΟΗΕ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πολύ απλό. Πώς εσείς αντιλαμβάνεστε τη σχέση μας με την Τουρκία τη στιγμή που θέλουμε να εντάξουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη και ταυτοχρόνως η Τουρκία βρίσκεται σε ενταξιακό καθεστώς που σας αφορά εσάς ως Επίτροπο. Και το δεύτερο ερώτημα. Ήρθε μήπως η ώρα να αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις μας καλής γειτονίας με επενδύσεις στις χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατήσουμε τον κόσμο αυτό στις χώρες του. Αυτά. And finally we go back to your home. Και γυρίζουμε στη δική σας χώρα, κύριε Επίτροπε, και στον κύριο Τσέγκα Ζάλαν από τον Κρυκό Εθνικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι η Ουγγαρία δεν έχει αλλάξει τη θέση σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική της διεύρυνσης. Θεωρεί πάντοτε ότι πρόκειται για μία από τις πιο στρατηγικής σημασίας πολιτικής ένωσης γιατί συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των ε, σημερών προκλήσεων της Ένωσης. Είναι πλέον προφανές ότι η πολιτική διεύνηση της Ένωσης έχει τελματώσει. Κατά την άποψή μας οι ανεπάρκειες στην πολιτική αυτή κυρίως προέρχονται από την αναξιόπιστη αυτή διαδικασία. Άρα ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θεσμικό ε, πλαίσιο. Ε, αν αυτό είναι το πρόβλημα ή αν πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτική βούλησης από τα κράτη-μέλη. Δεν είμαστε κατά της ενδεχόμενης ε, ανθεώρησης της διαδικασίας, αλλά αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία διεύρυνσης, παρακολύοντας την πρόοδο που αξίζουν οι χώρες αυτές. Τονίζουμε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης των ε, διαπραγματεύσεων με Σερβία και Μαυροβούνιο που έχουν ξεκινήσει ήδη. Κύριε Επίτροπε, πότε θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δύο αυτές χώρες, Σερβία και Μαυροβούνιο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Και τέλος, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω το λόγο σε έναν συνάλφο που διετέλεσε ευρωβουλευτής, αλλά τώρα έχει επιστρέψει στην εθνική πολιτική, τον κύριο Μάρκ Ντεμεσμάκερ. Καλώς ήρθατε Καλά είστε. Ναι, να μιλήσω ε, στα Ολλανδικά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που θα ήθελα να την είχα κάνει στον κύριο Μπορέλ, αλλά τέλος πάντων. Μπορώ και σε εσά, ε, κύριε Βαρχέλη, να αντιθέσω και έχει να κάνει με την ε, διεύρυνση και την υπεράσπιση των αξιών μας ουσιαστικά, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, της δημοκρατίας. Αυτά είναι η πεμπτουσία, είναι η βασική ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε και μια μεγάλη θική υποχρέωση και στη γειτονιά μας και στον υπόλοιπο κόσμο απέναντι Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε ένα κύρος και μια βαρύτητα όταν ε, και στην εξωτερική μας πολιτική και στην εσωτερική πολιτική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τα μέσα πολιτικής ε, όχι επιλεκτικά αλλά συλλογικά. Να μην κοιτάμε από την άλλη πλευρά όταν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ένωσης. Έχουμε μια επιλεκτική στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη, οι καταλανοί πολιτικοί διώκονται και αποστρέφουμε το βλέμμα. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε υπόψη. Δεν είναι μόνο η Ισπανία, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ε, και ο Ερτογάν είναι ένα παράδειγμα ε, που υποστηρίζει τη δίωξη Κούρδων πολιτικών και δίνει ως παράδειγμα προς μίμηση ε, τη δίωξη των καταλανών πολιτικών από την Ισπανία. Δεν θα πρέπει λοιπόν παντού να υπερασπιζόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, παντού ανά τον κόσμο. Δεν μπορεί να επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση εσωτερικά, στο εσωτερικό της, να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Γιατί τότε δεν ε, δίνουμε το σωστό μήνυμα, ούτε εντός ούτε εκτός. Πρόεδρος. Έχουμε τώρα την κυρία Χιμίνα την που και αυτή άφησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να πάει στο Εθνικό Κοινοβουλίο. Θέλω και εγώ να μιλήσω στα Ισπανικά. Για να πω και στον ε, προηγούμενο ε, συνάδελφο ότι στην Ισπανία καμία παραβίαση των δικαιωμάτων δεν υπήρξε. Και αν υπήρξε, τη διέπραξαν ακριβώς αυτοί που είναι φυλακοί. Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας τους καταδίκασε για ε, στάση, ε, και για προσπάθεια απόσχησης ε, και δια της βίας προσπαθούσαν, όχι μέσα σε ένα κοινοβούλιο όπως έπρεπε, όπως είναι το Ισπανικό Κοινοβούλιο, να το κάνουν. Γιατί το, ο Ισπανικό λαό έχει την κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει δια τη βία. Περί αυτού πρόκειται να το πω ξεκάθαρα. Στην Ισπανία δεν υπάρχει καμία έλλειψη ελευθερίας. Οι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι ε, πήραν αυτή την απόφαση, ε, την έτοιμη γορία αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ε, Ισπανία. Η Ισπανία υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί αυτοί που είναι στη φυλακή γιατί έκαναν ή θα μπορούσαν να είχαν κάνει πραξικόπημα σε ένα κοινοβούλιο όπως αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, αν είχαμε εγκληματίες, βουλευτές θα ήταν φυλακή. Επίτροπο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Τα προβλήματα που έχουν με τη Ρωσία συμπεριλαμβανομένη της κατοχής του εδάφους τους κατά πόσον θα ήταν πρόβλημα για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα πιστεύω όχι. Το έχουμε ήδη αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Το πρώτο στοιχείο βέβαια είναι η DCFTA. Μέσω της ε, συμμόρφωσης προς το 70% του ενωσιακού δικαίου μπορούν να ευθυγραμμιστούν σε κάθε πτυχή της ζωής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε και να τους βοηθούμε και αν δούμε και τα τμήματα ελευθέρων συναλλαγών των συμφωνιών αυτών, των FTA, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητα της ζωής της Ένωσης. Τώρα, αν έχουν πρόσθετες περιοχές όπου θα επιθυμούσαν στενότερη συνεργασία, με μεγάλη χαρά θα το κάναμε. Και στην περίπτωση της Ουκρανίας θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να τους διασυνδέσουμε πολύ πιο στενά υπό την έννοια των ψηφιακών ή άλλων υποδομών ή ενεργειακών υποδομών ή και μεταφορικών. Υπάρχουν κάποια πράγματα δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που και εκείνοι θα ήταν έτοιμοι να κάνουν. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο εμπόδιο λόγο της κατοχής εδάφους τους. Αντίθετα, εμείς πρέπει ακόμα περισσότερο να συνεργαζόμαστε μαζί με τις χώρες αυτές καθότι βρίσκονται υποπίεση από τη Ρωσία. Τώρα για το ρόλο των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Εχθές το συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και το μήνυμα είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε άπαντες να επανέλθουν στα Εθνικά Κοινοβούλια και να δρουν πολιτικά εκεί θα ενθάρρυνα άπαντες να επανέλθουν στα Εθνικά Κοινοβούλια και να κάνουν κάθε προσπάθεια από εκεί. Διαφορετικά οι χώρες αυτές δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας πείσουν, να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι μπορούν να συμμετάσχουν ως πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειαζόμαστε ένα κοινό ελάχιστο παρανομαστή, εθνικός μιλώντας, για την ενταξιακή διαδικασία. Πρέπει να συμφωνήσουμε για θέματα που άπτονται της δικής τους συμμετοχής ή ένταξης. Θα ενθάρρυνα όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να δράσουν κατά τον τρόπο αυτόν. Μόνος μου δεν πρόκειται να καταφέρω τίποτε τέτοιο. Εγώ ήδη ζήτησα τη βοήθεια της Επιτροπής σας και θα συνεχίσω να το κάνω. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ακούν αλλήλους ίσως περισσότερο από ότι οποιονδήποτε άλλον. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Εγώ πιστεύω ότι τα μέλη του οίκου αυτού ε, βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κεντρική θέση να ε, ε, εξηγήσουν σε όλους γιατί είναι τόσο κρίσιμη σημασία στα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ θα βοηθήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουν να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Γιατί έχουμε πολλά να πετύχουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, νομίζω ότι εξυπακούεται ότι η παρουσία μας ε, ως προς τις δημόσιες σχέσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Για να το πω έτσι. Και κοιτώντας τα μεγέθη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της που κάνουν τα περισσότερα για τις χώρες της περιοχής. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί υπό την έννοια της εικόνας μας ή των δημοσίων σχέσεών μας έχουμε τόσο ελλειπή αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή που κάνουμε στην Ουκρανία, με το EU for You, για να εξηγήσουμε καλύτερα στους πολίτες των χωρών τι κάνουμε και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Υπάρχει και ένα άλλο βέβαια ουσιώδος θέμα, ότι οι πράξεις μας, οι δράσεις μας είναι διαρρεμένες σε διάφορες μικρές ομάδες, αντί να εστιαζόμαστε σε πιο μεγάλα έργα, μεγαλύτερα οράματα, μεγαλύτερου αντικτύπου και πιο εμφανή. Αυτές είναι οι δύο προσεγγίσεις που εξετάζω Αλλά ως προς την διαδικασία της διεύρυνσης, αυτή η διάσταση θα είναι πολύ σημαντική, πιστεύω. Επί της Τουρκίας τώρα. Η προσέγγιση μας νομίζω είναι σαφής για την Τουρκία. Έχουμε ουσιαστικότατα προβλήματα στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Με τις παράνομες ε, εξορίξεις έξω από την Κύπρο. Το Συμβούλιο έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί σχετικά με την πιθανότητα κυρώσεων. Δεν υπάρχει αλλαγή στην γραμμή αυτή. Θα συνεχίσουμε με χρυσό του εγκαταλείψουν τη δραστηριότητα εξορίξεων, την παράνομη δραστηριότητα. Επίσης, για τις διαπραγματεύσεις ξανά και ξανά έχουμε θέσει τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ελευθερία τύπου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κράτηση δημοσιογράφων, ε, διάφορα κρούσματα που είναι υποχωρήσεις ως προς το κράτος δικαίου. Αυτά είναι πραγματικές ανησυχίες και πρέπει να τα εξετάζομαι όσο η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της υποψήφια χώρα είναι από την άλλη μεριά η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του στα θέματα μετανάστευση και επομένω πρέπει κανεί να ξαναδεί το θέμα των σχέσεων με τη χώρα αυτή συνολικά. Θα πρέπει να, δει, να γίνει αυτό και εδώ, στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Και πρέπει να δούμε τις αδυναμίες, αλλά για τα ισχυρά μας σημεία σε αυτή την προσέγγιση. Για τη Σερβία και το, Μοντενέ, ή το Μαυροβούνιο, με Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν δίνοντας τους κίνητρα να μας πλησιάσουν το συντομότερο δυνατόν. γιατί με το παράδειγμα της οικονομίας της αγοράς μόνο μέσω αυτού μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί είναι θεμελιώδες να υπάρχει δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελευθερία τύπου. Γιατί αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά χωρίς τα οποία το επιχειρήν δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα. Χρειαζόμαστε μια οικονομία της αγοράς που να βασίζεται στο κράτος δικαίου και που να είναι καλή και για μας και για εκείνους. Αυτό θα νομίζω ότι θα τους επιτρέψει ταχύτερα να καλύψουν το έδαφος. Νομίζω ότι έχω απαντήσει, Πρόεδρε, τις ερωτήσεις. Και άλλο γύρο θέλετε, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Ε, τελικό, τελευταίος γύρος. Μόνο με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων πριν από αυτό όμως, Επίτροπε, εγώ ήθελα ένα σημείο να πω σχετικά με τις ε, γεωτρήσεις στα Κυπριακά Ήδατα. Είχαμε συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Χαιρετήσαμε το, τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου για τα μέτρα που θα αναλάμβανε, αλλά τώρα περιμένουμε να υλοποιηθούν κυρώσεις με απαγορεύσεις ταξιδίων και παγώματα περιουσιακών στοιχείων για τους υπευθύνους. Γιατί μόνο τότε θα μας πάνουν στα σοβαρά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάω τώρα στον τελευταίο γύρο. Ο κύριος Πετρουτσέλη από την Ιταλία δεν είναι εδώ, μάλιστα. Ο κύριος Μπίγνιεφ από την Πολωνία, παρακαλώ. Please. Okay, thank you, thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι μια αποτυχία έναρξη τη διαδικασίας προσχώρησης στα Δυτικά Βαλκάνια συμβαδίζει με την αποτυχία του να δημιουργήσουμε καλών διάβλων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων προκειμένου να εξηγηθεί η κατάσταση στους πολίτες επιτόπου. Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτό και λογικό να περιγράψουμε το χρονοδιάγραμμα για την ε, μελλοντική διαδικασία προσχώρησης για να είναι πιο ενθαρρυντικά τα πράγματα για αυτές τις δύο χώρες, ότι δεν θα διαρκέσει δεκαετίες η διαδικασία, αλλά κάποια λίγα χρόνια. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Μπορείτε παρακαλώ αν έχετε συζητήσεις ε, να τη συνεχίσετε εκτός της αιθούσης. Αναφέρομαι στους Γερμανούς συναδέλφους. Επόμενος ομιλητής από τα κάτω χώρες, ο κύριος Δίτριχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθώς ε, πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος σύντομα, αλλά θα εξακολουθήσει να είναι η γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Επίτροπε, να δούμε πέρα από το Brexit και παραδείγματο χάρη σε πέντε χρόνια. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ζουρτάν, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, είναι πολύ σημαντική η ε, πολιτική της γειτονία και της ανατολικής εταιρική σχέσης και η πολιτική της διεύρυνσης στις χώρες της Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ζωτική σημασία. Ε, τα επίμαχα σημεία που είχαμε την τελευταία εβδομάδα απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία μας δείχνουν την αλήθεια του θέματος. Μπορείτε, κύριε Επίτροπε, να μας πείτε ποια είναι η ανάλυση σας για τη διάρθρωση μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και της πολιτικής διεύρυνσης. Δεύτερη ερώτηση. Το προηγούμενο Σεπτέμβριο η τελική δήλωση της Συμπροεδρίας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΑ και για την ΚΠΑ ε, ε, υπέγραφε ότι η διαδικασία εσωτερική μεταρρύθμιση και προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συμβαδίζουν για να ενισχυθούν. Πώ ε, ε, εσείς αντιλαμβάνεστε το σύνδεσμο μεταξύ πολιτικής διεύρεσης και της εσωτερικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημητρέσκου από τη Ρουμανία. Δύο ερωτήσεις ε, θέλω να σας θέσω. Καταρχήν θα ήθελα την άποψή σας για τη Μολδαβία σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση και λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική κατάσταση που έχουμε τώρα στην Μολδαβία, δηλαδή ότι η κυρία Μαγιασάντου έχασε την κυβέρνηση. Επίσης, Σήμερα αλλά και τις τελευταίες μέρες μιλήσαμε ιδιαίτερα για την αναγκαιότητα που προτείνουν κάποιες χώρες, κυρίως η Γαλλία, να υπάρχουν οι κανόνες για την διαπραγματευτική διαδικασία, για την πολιτική διεύρυνση. Οι τελευταίες 13 ε, χώρες μπήκαν στην Ένωση σεβόμενες τα κριτήρια της Κοπενχάγης. και ακολούθησαν διαπραγματευτική διαδικασία σε κάθε κεφάλαιο. Αν χρειάζεται να έχουμε νέους κανόνες, εντάξει, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε κάποια ιδέα σχετικά και αν έχετε κάποια ιδέα αν πρόκειται για τους όρους, δηλαδή με αυστηρούς κανόνες και με προθεσμίες, γιατί για τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα απέναντι στη διαδικασία. Και καλή επιτυχία για τη θητεία σας. Ευχαριστούμε. Να σας ενημερώσω ότι η κυρία Μαγιά Σάντου θα έρθει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο για να μας ενημερώσει για την κατάσταση στη Μολδαβία. τελευταίος, από την Τσεχική Δημοκρατία, ο κύριος Μπένεσικ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θέλω να υποστηρίξω τόσο υπόθηκαν εδώ. Οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να έχουν προοπτική. Γιατί αν εμεί αφήσουμε το κενό, κάποιο άλλο θα το καταλάβει. Και αυτό δεν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε συμφέρει τι χώρε αυτέ. Να καλύψει κάποιο άλλο το κενό. Και είχε πει ο Επίτροπος Χάν, αν δεν φέρουμε σταθερότητα στα Βαλκάνια, τα Βαλκάνια θα φέρουν αστάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση για την ανατολική εταιρική σχέση. Πολλά υπόθηκαν, αλλά ως εκπρόσωπος της Τσεχικής Δημοκρατίας ε, η οποία συνέβαλε στη γένεση της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πριν 10 έτη. Θέλω να ρωτήσω αν ε, σκοπεύετε να προβείτε σε σοβαρές αλλαγές στη φιλοσοφία, γιατί έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση τελευταία. Έχουμε εξελίξει σε διάφορες χώρες. Αυτή είναι λοιπόν η συγκεκριμένη ερώτηση που σας θέτω. Σχεδιάζετε κάποιες πιο σοβαρές αλλαγές στην προσέγγιση στην ανατολική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Και τέλος, ο κύριος Μουλίτεν Γιωκάνοβιτς από το Μαυροβούνιο, από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απευθυνθώ. Προέρχομαι από το Μαυροβούνιο. Ανήκω στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Χτες συμμετείχα σε μια συνεδρίαση για την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια άποψη. Ακούσαμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη κριτική της νέας μεθοδολογίας που προτείνεται από τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά δεν ε, συμμεριζόμαστε όλοι την άποψη αυτή. Κάποιοι θα την υποστήριζαν, γιατί οι πολίτες ε, θα ήταν οι πρώτοι που θα ένιωθαν ε, κάποια ωφέλη της διαδικασίας προσχώρησης. Μέχρι τώρα ε, οι πολίτες δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ποια είναι τα ωφέλη της διαδικασίας διεύνησης. Και θέλω να ρωτήσω, δεν θα ήταν λογικό οι ευρωπαϊκές αξίες να ε, μπορούν να προβάλλονται καλύτερα στα Δυτικά Βαλκάνια και να υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Ακόμη και αυτή η ιδέα κρίση μικρής Σέγγεν φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ενθαρρύνετε το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία Βαρζεγοβίνη να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία και ότι θα πρέπει μάλιστα να καταργήσουμε και τα σύνορα μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, κατόπιν η ολοκλήρωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι λιγότερο προβληματική. Η ένταξή μας θα είναι λιγότερο προβληματική, γιατί ε, ε φυσικά ε, δεν είναι φυσικό να θέλουμε ε, να έχουμε μεγαλύτερο κλείσιμο με την Δανία, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε τα σύνορα με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, παραδείγματο χάρη. Σα ευχαριστώ. Και βάσει των όσων είπατε, Δευτέρα Τρίτη ήμουν στο Βελιγράδι και όπως πολλοί από εμά ε, που ταξίδευσαν στα Δυτικά Βαλκάνια, το πρώτο βήμα ολοκλήρωση που όλοι θα κλεισορίσουμε είναι να καταργήσουμε τα τέλη περιαγωγή. Είναι απίστευτο ότι περνά τα σύνορα και ξαφνικά ε, είσαι σε εντελώ διαφορετικό καθεστώ σε σχέση με την τεχνολογία των κινητών. Και φυσικά να καταργούμε οποιαδήποτε σύνορα πάντα βοηθά στα Δυτικά Βαλκάνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω κάλυψα όλα τα αιτήματα ήταν πολύ μακρύς ο κατάλογο και έχουμε τώρα την τελευταία ε, απάντηση από τον Επιτροπό Λιβέρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις αφορούσαν το χρονοδιάγραμμα της διεύρυνσης. Ε, Ακαμφθόδες το ερώτημα. Μπορεί κανείς να πει έτσι κάπως απερίσκεπτα 2025, αλλά τα έχουμε πει και ξαναπεί. Το έχουμε δει αυτό το έργο. Το θέμα είναι η διαδικασία που θα υιοθετηθεί να μπορέσει να φέρει σε αίσιο πέρας την διεύρυνση προς αυτές τις χώρες. Εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτή την πενταετία και τα σχέδιά μου είναι στο πέρας της πενταετίας αυτής τουλάχιστον μία χώρα να είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορώ να σας πω. Στο τεφαρτό χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάτι περισσότερο, αλλά με τα χαρά μπορώ να το κάνω ε, αυτό που σας είπα, να δεσμευτώ ως προς αυτό τουλάχιστον. Τώρα, για το ερώτημα κατά πόσον η διεύρυνση και η εμβάθυνση εξαρτώνται η μία από την άλλη. Ε, δεν το νομίζω. Νομίζω ότι η διεύθυνση είναι δυνατή χωρίς μίζωνα θεσμική αναδιάρθρωση. Αν συμφωνήσουμε πάνω σε μια ε, θεσμική αναθεώρηση, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι όμως ε, προϋπόθεση αυτή καθεαυτή για μια διεύρυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με 28 κράτη για μια ακόμη φορά. Θα πρέπει να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει με άλλο ένα κράτος. Αν ένα μήνυ Σέγγεν θα ήταν καλή ιδέα, ακούστε οποιαδήποτε περιφερειακή συνεργασία πριν την προσχώρηση μεταξύ χωρών Δυτικών Βαλκανίων, είναι κάτι καλοδεχούμε. Ένα μήνυ Σέγγεν εμένα ε, φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Με μια προϋπόθεση όμως, ότι θα πρέπει όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν, να είναι ανοιχτό προς όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, και να πω εγώ ότι με βρίσκει σύμφωνο, ε, σίγουρα θα μπορέσει να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων, τι εμπορικέ συναλλαγέ, τι διαπροσωπικέ επαφέ. Οφέλη μπορεί να φέρει, άρα εγώ το επικροτώ κάτι τέτοιο, όμω, θα έλεγα ότι καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσχωρήσουν, τη βέβαια. Για τη Μολδαβία και την κατάσταση στη χώρα αυτή, εμεί ε, πολύ κοντά, από πολύ κοντά παρακολουθούμε την κατάσταση και βλέπουμε ότι είναι κάπως απρόβλεπτη η τωρινή πολιτική κατάσταση, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον. Η δική μας γραμμή δεν έχει αλλάξει. Θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση της Μολδαβίας. Όσο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις και θα συνεχίσουμε να βοηθούμε και οικονομικά και θεσμικά τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Σε διαφορετική περίπτωση, για μια ακόμη φορά, θα πρέπει να ανασταλεί χρηματοδότηση ή να αληφθούν άλλα μέτρα. Άρα πρέπει να παραμείνει σε τροχιά η Μολδαβία. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί αυτό. αν προβλέπετε διεύρυνση προς τη Μολδαβία. Ακούστε προς το παρόν, δύσκολο, πολύ δύσκολο το βλέπω να δοθεί η προοπτική διεύρυνση. Αλλά από ό,τι ξέρω και το είπα ήδη, είναι ότι η DCFTA, η συμφωνία αυτή για τις ελεύθερες προβλέπει ε, πολλά περιθώρια βελτίωση των αντιμετωπιστικών σχέσεων και όταν θα έχουμε εφαρμόσει αυτή την ε, συνολική συμφωνία, τότε θα έχουμε εντοπίσει ε, τις δυνατότητες ε, ε, για οποιοδήποτε άλλο τομέα συνεργασίας. Ούτως ή άλλως οποιαδήποτε χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη. Αυτό είναι μια διαφορετική διαδικασία. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά την ανατολική γειτονία και τα μελλοντικά μας σχέδια, είμαστε μέσω περίοδου προβληματισμού. Δεν ξέρω ακριβώς τι νέες ιδέες θα προκύψουν. Αλλά μπορώ να σας πω ήδη κάτι. Και αυτό είναι το εξής. Προσέγγιση. Οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο βαθιάς συνεργασίας, θα περιληφθεί σε αυτή τη στρατηγική, αλλά είναι πολύ νωρίς. Να πει κανεί ε, τι άλλα νέα στοιχεία θα μπορούσε κανεί να αναμένει από εμά. Ολοκληρώνει το που να είναι η δημόσια διαβούλευση, μετά θα γίνει εσωτερικά μια διαβούλευση και θα έρθουν σε επαφή με τις χώρες και με τα κράτη-μέλη βέβαια, τα οποία και θα ενημερώσουν. Θα ζητήσουμε τη γνώμη σου πριν κατάληξουμε τις προτάσεις μας. Τι άφησα για τελευταίο. Το κερασάκι στην τούρτα άφησα. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Αστείο είναι έτσι, με το πάρτε σοβαρά θα μπορούσαμε να έχουμε δυτική εταιρική σχέση ε, με τη Βρετανία, αν το επιθυμεί και υπό και προϋποθέσεις βεβαίως. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να δούμε τι θέλει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θέλει αυτό να είναι η μελλοντική μας σχέση. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο κάποιου άλλου. Και όταν ο κάποιο άλλο αυτό έχει πλέον καθορίσει το πλαίσιο των ερωτικών σχέσεων, θα πάρω ίσω εγώ το χαρτοφυλάκιο. Αλλά ο προηγούμενο επίτροπο, ο Μισελ Μπαρνιέ, ε, είναι ο αρμόδιο ε, και αυτόν πρέπει να ρωτήσετε. Το λιγότερο πάντως ε, που είναι απαραίτητο είναι μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ε, αλλά θα σας τα πει πολύ καλύτερα ο Μισελ Μπαρνί από μένα. Ευχαριστώ πρόεδρος, αγαπητοί συνάλφοι. Πριν σηκωθείτε να φύγετε, επιτρέψατε μου να κήρυξω τη λήξη αυτής της συνεδρίασης, ευχαριστώντα πρώτα απ' όλα τον ε, Επίτροπο Βαρχέλη για τον πολύ χρόνο που μας διέθεσε, πατώντας και σε όλα τα ερωτήματα. Και ε, σε αυτό το ε, πολύ μικρό χρονικό διάστημα βλέπω ότι έχετε εξοικειωθεί ε, με πολλά θέματα. Έχετε έτσι ήδη μελετήσει ενδελεχώς την πολιτική κατάσταση σε πολλές χώρες. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια που διοργάνωσε μια εξαιρετική συνάντηση. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστήσω προ του συναδέλφου μα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους συνεργάτες σας. Ήρθατε εδώ, μας ε, ε, δώσατε και τις δικές σας απόψεις. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες οι ανταλλαγές αυτές και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι αν ε, συμφωνείτε. Επόμενη συνάντηση λοιπόν στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για την ΚΕΠΑ, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική Πολιτική Ασφάλειας, 2 με 4 Μαρτίου στο Ζάγκρεμπ, Υπουργό Εξωτερικών τη Κροατία. θα συζητήσουμε το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζουμε για εσά ε, σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο απόγευμα εδώ στις Βρυξέλλες. Καλή επάνδρωση στις χώρες σας ε, και θα τα ξαναπούμε το Μάρτιο στο Ζάγκρεπ. Πέρα στη συνεδρίαση. Tök jó olyan témákról esett szó, amit még jól